Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Πλησιάζουμε όλο και περισσότερο στις καλοκαιρινές διακοπές. Το γνωρίζω. Και αυτό είναι πολύ καλό νέο. Και άλλωστε μπορούμε και να το διαπιστώσουμε, γιατί η Επιτροπή μας δεν φαίνεται καν να είναι Επιτροπή ΛΥΜΠΕ δεν μοιάζει καθόλου με τη συνηθισμένη προσέλευση που έχουμε συνηθίσει. Έχουμε λοιπόν φτάσει στην τελική ευθεία αγαπητοί συνάδελφοι και είμαστε στο σημείο 17. Συζητούμε για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο και το πρόγραμμα εργασίας αυτής για το 2011 και είναι εδώ ο εκτελεστικός διευθυντής, ο δόκτωρ Ρόμπερτ Βίσερ, τον οποίο θερμότατα καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε στην απογευματινή συνεδρία της Επιτροπής μας. Με μεγάλη χαρά αναμένουμε την έναρξη λειτουργίας αυτής ε, της νέας ε, υπηρεσίας υποστήριξης για το άσυλο και με πολύ χαρά θα ακούσουμε και το πρόγραμμα εργασίας για το 2011. Απλώς να σας υπενθυμίσω ότι αυτή η νέα ευρωπαϊκή υπηρεσία εγκρίθηκε στη Βαλέτα της Μάλτας, εγγενιάστηκε στις 19 Ιουνίου με σκοπό να υποστηρίξει το κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου που είναι ένα από τα συστατικά στοιχεία, για να το πω έτσι, της φιλοδοξίας του ευρωπαϊκού χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα στο πλαίσιο της συνθήκης της Λισαβόνας. Οπότε, καλωσορίζουμε τον κύριο Βίσερ και μετά θα έχουμε και τη συζήτηση μαζί του. Κύριε Βίσερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να είμαι εδώ ενώπιον σας και πάλι στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών από τις 9 Δεκεμβρίου πέρσι που είχα την ευκαιρία να αυτοπαρουσιαστώ υποψήφιος για αυτό το αξίωμα ενώπιόν σας και μετά διορίστηκα σε αυτό το αξίωμα από την 1η Φεβρουαρίου 2011, εφέτος δηλαδή. Και χαίρομαι τώρα που μπορώ να σας παρουσιάσω το πρόγραμμα εργασίας μας για το 2011 που έχει διανεμηθεί προηγούμενα σε εσά. Από τότε συνέβησαν κάποια συμβάντα και δραστηριότητες που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν για την κατάσταση παράδειγμα στη Μεσόγειο υπάρχουν κάποιες μεταθέσεις προτεραιοτήτων αλλά σε μεγάλο βαθμό βρισκόμαστε ευθυγραμμισμένοι με το πρόγραμμα όπως ε, υποβλήθηκε. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό επικεντρώνεται στις προτεραιότητες που παρουσιάζονται όσον αφορά τον κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το πρόγραμμα για τη Στοκχόλμη και το πρόγραμμα δράσης για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Επιτρέψτε μου πολύ σύντομα να επισημάνω κάποια από τα στοιχεία αυτού του προγράμματος εργασίας. Πρώτα απ' όλα φυσικά, ξεκινώντας με την οργάνωση από μηδενικού σημείου, ο πρώτος απασχολούμενος σε αυτόν τον οργανισμό που ήμουνα, δηλαδή πρόσληψη, χρηματοδότηση, προκηρύξεις και υποβολή προσφορών και στην διαδικασία στελέχωσης αυτή του οργανισμού μας. Τώρα έχουμε συνεντεύξεις με ένα μεγάλο αριθμό υποψηφίων για 27 μόνιμα στελέχη και για αυτές έχουμε 2.500 υποψηφίους για αυτές τις 27 θέσεις. Έχουμε πολλούς λοιπόν, πολλή δουλειά, αλλά με την υποστήριξη της Επιτροπής θα καταφέρουμε να τα βγάλουμε πέρα. Θα πάει όμως κάποιο χρόνο όλο αυτό διαδικαστικά. Δεύτερον, χρησιμοποίησα τους ε, όπως αποκαλούμε επικουρικούς ε, εθνικούς εμπειρογνώμονες 11 ή 12 συνολικά για φέτος οι περισσότεροι από τους οποίους έχουν ήδη διοριστεί κατά τα τέλη του 2011 ελπίζω να λειτουργούν και να έχουν προσληφθεί 40 στελέχη που θα απασχολούνται στον οργανισμό μας. Ταυτόχρονα όταν ανέλαβα το αξίωμά μου ζητήθηκε και έπρεπε να δώσουμε πλήρη υποστήριξη για την κατάσταση των μεταναστών στην Ελλάδα και χάρη στις πρωτοβουλίες και την πραγματογνωμοσύνη κάποιων κρατών μελών και χάρη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ύπατη αρμοστία για τους πρόσφυγες των Ηνωμένων Εθνών καταφέραμε να εκπονήσουμε τις λεπτομέρειες των δράσεων για τους πρόσφυγες και μετανάστες στην Ελλάδα και στις αρχέ Φεβρουαρίου αποκοινούμε τον Έλληνα Υπουργό κύριο Παπουτσί μπόρεσα να υπογράψω το λειτουργικό πρόγραμμα και τις, οι πρώτες ομάδες αμέσως μετά ε, στάλθηκαν, ε, επικουρικές ομάδες για το άσυλο στην Ελλάδα. Χαίρομαι που καταφέραμε από κοινού με την Ελλάδα να δρομολογήσουμε όλες αυτές τις δράσεις σε αυτό το πλαίσιο. Και μέχρι σήμερα η δουλειά πραγματικά προοδεύει ανάλογα σύμφωνα με το πρόγραμμά μας και προοδεύει και προχωρά σύμφωνα με το σχέδιό μας. Σημαντικό τώρα είναι για την κατάσταση στην Ελλάδα και η βελτίωση που πρέπει να σημειωθεί. Επίσης είναι σημαντικό το πρόγραμμα να έχει τέτοια μορφή ώστε μια σταθερότερη, διαρκέστερη κατάσταση αναβαθμισμένης ε, λειτουργίας να μπορέσει να κατάρτιστεί, να λειτουργήσει και για τα θέματα ασύλου και για τα θέματα υποδοχής. Πέρα από το πρόγραμμα για την Ελλάδα και την υποστήριξη, ξεκινήσαμε και άλλες δραστηριότητες. Πιο συγκεκριμένα μπορώ να επισημάνω το πρόγραμμα για το Ευρωπαϊκό Ασύλο και την κατάρτιση για το Ευρωπαϊκό Ασύλο, ένα σύστημα κατάρτισης. Και από το Σεπτέμβριο 2011 θα ξεκινήσουμε με τη διοργάνωση αυτών των σεμιναρίων κατάρτισης. Δεύτερο σημαντικό ζήτημα, το οποίο αξίζει να τύχει μεγάλης προσοχής, είναι οι πληροφορίες για την χώρα προέλευσης. η ιστοσελίδα, ο ιστότοπος σε σχέση με αυτά τα στοιχεία, ώστε να μπορούν να, έχουν πρόσβαση τα κράτη-μέλη σε σχέση με αυτά τα στοιχεία. Θα έχουμε την εκκίνηση φέτος και ε, το ΙΑΣΟ θα αναλάβει μετά την ε, ευθύνη για όλα αυτά. Το πρόγραμμα αυτό μέχρι τα μέσα του επόμενου έτους θα έχει οδηγήσει σε κοινή έκθεση για τις χώρες προέλευσης, κυρίως για τη χώρα προέλευσης Αφγανιστάν. Τρίτον, δώσαμε προσοχή, δίνουμε προσοχή στην υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δράσης για τους μη συνοδευόμενους ανήλικους. Κατά το δεύτερο ήμιση αυτού του έτους θα πρέπει να ξεκινήσει στη λειτουργία του. Με συμμετοχή επίσης και της Frontex. Τέταρτος άξονας. Η δυνατότητα παρέμβασης όσον αφορά το Asylum Intervention Pool υποστήριξη όσον αφορά για την ανακούφιση συγκεκριμένων πιέσεων έχουμε περίπου 350 πραγματογνώμονες που έχουν προσθέσει τα ονόματά τους σε αυτές τις ομάδες, σε αυτό το ε, όργανο. Και όπως είπαμε για την κοινωνία των πολιτών και την ε, δράση και εμπλοκή όσον αφορά τα θέματα ασύλου και μετανάστευσης θα έχουμε ένα πρώτο φόρουμ, ένα σεμινάριο με την κοινωνία των πολιτών αλλά με επίσης πανεπιστημιακούς, ακαδημαϊκούς εκπροσώπους ε, ώστε να μπορέσουμε να δραχθούμε τις ευκαιρίες και να εκμεταλλευτούμε την πείρα που, έχει, ε, που έχουν οι εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών για αυτά τα θέματα. Όπως προανέφερε ο Πρόεδρος στις 19 Ιουνίου η επίσημη τυπική ε, έναρξη σε σχέση με τη Μάλτα και η έδρα όσον αφορά την Μάλτα καθώς επίσης ε, και οι συμβάσεις ε, για τη στέγασή μας στην πρωτεύουσα της Μάλτας όλα αυτά λειτουργούν και ξεκίνησαν μέχρι σήμερα αντιμετωπίζουμε Πρόεδρε μεγάλες προσδοκίες που πρέπει να ανταποκριθούμε σε αυτές Πήγα πρόσφατα τις, τελευταίε τελευταίες μέρες στη Βαρσοβία σε σχέση με την ε, διάσκεψη που είχαμε για την κοινή πολιτική, ευρωπαϊκή πολιτική για το άσυλο. Ήταν επαρκώς σαφές ότι θα πρέπει να ενταχθεί αυτό το θέμα ως προοπτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα κοινό ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου. Όμως, τους τελευταίους μήνες είναι σαφές πλέον ότι η απάντηση μπορεί να λειτουργήσει αν θα έχουμε την αναγκαία υποστήριξη, υποστήριξη των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά επίσης και σε μεγάλο βαθμό εξαρτώμαστε από αυτή την υποστήριξη, την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μέχρι τώρα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση σημειώνω ότι υπάρχει η δέσμευση η εμπλοκή σας να μας ε, επικουρείτε και να μας συνδράμετε. Τώρα, <clears throat> Δύο λόγια για τη συνέχιση του προγράμματος ε, για το 2012. Οι ίδιες δραστηριότητες θα πρέπει περαιτέρω να αναπτυχθούν. Πέρα από αυτά θα επικεντρωθούμε στην ε, μεταγκατάσταση ε, προσφύγων και μεταναστών όσον αφορά και τις εξειδικευμένες εκθέσεις των χωρών προέλευσης. Υπάρχουν πολύ μεγάλες προσδοκίες, Πρόεδρε. Βλέπω μηδενική σημαντικό ποσοστό αύξηση του προϋπολογισμού ισχύει επίση και για την ΙΑΣΟ. Έχουμε μείωση κονδυλίων κατά περίπου 20% για έναν οργανισμό που δεν έχει καν το ελάχιστο δυναμικό να αντιμετωπίσει μια δυσχερέστατη κατάσταση. Όλα αυτά θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Με χαρά σας παρουσιάζω το πρόγραμμα εργασίας μα. Πολλή δουλειά έχει επενδυθεί σε αυτό και πρέπει να συνεχιστεί. Σα ευχαριστώ πολύ. Και εμεί σα ευχαριστούμε. Να είστε βέβαιος ότι εμείς σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία και σε εσά ε, και στο ΕΑΣΟ, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο. Σας ευχόμαστε και σας προσωπικά κάθε επιτυχία ως επικεφαλής της ε, συγκεκριμένης υπηρεσίας υποστήριξης. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ρωτήσω τους εκπροσώπους Ευρωπαϊκής Επιτροπής αν θέλουν να πάρουν το λόγο. Αν όχι, τότε να αρχίσουμε τη συζήτηση με τον κύριο Κάμπ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αν είναι παρόν ο κύριος Φίσερ, κάποιες αναμνήσεις από τα νιάτα μας έχουμε και από το Ολλανδικό Κοινοβούλιο είχαμε επαφή με τον κύριο Φίσερ. Αυτή η ιστορία λοιπόν αυτό, το, αυτό μπορεί να τύχει συνέχεια σας σίγουρα. Πρώτον σας ευχαριστώ πολύ για την εισήγησή σας και για το σαφές κείμενο όσον αφορά το πρόγραμμα εργασίας σας. Θα είχα αμέσως τέσσερις ερωτήσεις ε, να διατυπώσω βρισκόμαστε στην εναρκτήρια, στην αρχική φάση αυτού του κοινοτικού εγχειρήματος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Υποστήριξης για θέματα ασύλου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορούσε, δεν κατάφερε να δραστηριοποιηθεί αυτή η υπηρεσία. Οι Ευρωπαίοι πολίτες θέλουν να δουν πράξεις, χειροπιαστά αποτελέσματα από αυτό το, τον οργανισμό, από αυτό τον φορέα και με τη συμμετοχή όσον αφορά ε, θα δείτε ότι είναι σημαντικό το θέμα αυτό και πρέπει να ληφθεί υπόψη. Έχω το εξή ερώτημα. Αφορά την αποτελεσματικότητα του προγράμματος για την Ελλάδα. Είπατε ότι κάποιοι επαΐοντες πήγαν εκεί και κάτι έγινε. Τώρα τι έγινε. Έκλεισαν τα σύνορα προς την Τουρκία. Είναι στεγανά πλέον. Οι Έλληνες έχουν και είχαν πολλά προβλήματα και σε άλλα επίπεδα. Το γνωρίζουμε αυτό. Ποια αποτελέσματα χειρόπιαστα μπορείτε να μας αναφέρετε σε σχέση με το burden sharing, τον επιμερισμό βαρών και καθηκόντων. Ποια επιτυχία και ποια αποτελέσματα είχε χειροπιαστά το πρόγραμμα υποστήριξης για την Ελλάδα. Δεύτερον, πότε <clears throat> θα είχε ολοκληρωθεί αυτή η αρχική φάση λειτουργίας. Πότε θεωρείτε ότι θα έχετε φτάσει στο ρυθμό, ας το πω έτσι, πορείας κανονικής ε, λειτουργίας σας. Πόσο καιρός θα χρειαστεί για να φτάσετε στον κανονικό ρυθμό λειτουργίας σας. Τρίτη ερώτηση. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που ήδη τώρα, σήμερα, λαμβάνουν υπόψη όλα αυτά τα οποία κάνετε και όσον αφορά τις δράσεις, για παράδειγμα τα συμβάντα μεταξύ Ιταλίας-Γαλλίας, όσον αφορά τους τινήσιους πρόσφυγες που ε, επισκέφθηκαν την Ιταλία και ήθελαν να συνεχίσουν μετά στην Γαλλία και σταμάτησαν οι Γάλλοι αυτούς στα σύνορα, δεν είναι ακριβώς ένα πρότυπο επίλυσης προβλημάτων. Τι γίνεται ακριβώς. Ο κύριος Σαρκοζή θυμώνει όταν φταρνιστεί κάποιος, έτσι δεν είναι. Τι γίνεται λοιπόν με αυτά τα θέματα. Και τελευταία ερώτηση για το burden sharing, τον επιμερισμό βαρών και καθηκόντων. Τι, πώς προχωράει το θέμα αυτού του επιμερισμού καθηκόντων και βαρών. Δηλαδή κάποιοι σε άσυλο πηγαίνουν παραπέρα, προωθούνται παραπέρα χωρίς κάποιες ε, δοκιμασίες ή ε, ε, κάποιες εξετάσεις ή γίνονται κάποιες εξετάσεις και μετά γίνεται η περαιτέρω μετάθεσή τους, μεταγκατάστασή τους. Τι γίνεται ακριβώς και ποιες εξελίξεις προβλέπετε τα επόμενα χρόνια. Σας ευχαριστώ. Thank you. Thank you. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Η κυρία Σίπερ. Σας ευχαριστώ πολύ. Δυστυχώς έχουμε περιορισμένο χρόνο, διότι θα ήθελα κάποια συγκεκριμένα πράγματα να μάθω. Η δική σας επιτροπή είναι μια μεικτή επιτροπή με σταθερά στελέχη και με την χρήση ε, επικουρικών υπαλλήλων από τους εθνικούς επαΐοντες. Θα με ενδιέφερε αυτή η συνεργασία αυτών των τελείως διαφορετικών ανθρώπων να μάθω πώς λειτουργεί και πώς αυτοί οι επαΐοντες, π.χ. για παράδειγμα στην Ελλάδα, στην Ελλάδα από τη Γερμανία οι αποσταλμένοι θα μπορούσαν στην Ελλάδα να συμμετέχουν. Η Ελλάδα σε πολλές πτυχές, πολυσχηδώς, είναι μια δύσκολη περίπτωση χώρας. Η Ελλάδα θα πρέπει να εξοικονομήσει, εξοικονομήσει όλο λιτότητα και μ, περιστολή δαπανών και όταν γίνονται τέτοιες περιστολές και τέτοια λιτότητα διαρωτάται κανείς τι μπορεί να επιτευχθεί, μπορεί κάτι να γίνει για να βελτιωθεί η κατάσταση στην Ελλάδα και πώς είναι η συγκεκριμένη υποστήριξη του γραφείου σας, της δικής σας υπηρεσίας προς μια τέτοια χώρα όπως την Ελλάδα, ώστε να συνοδεύσετε επικουρικά τις δράσεις σας. Και το θέμα των ασυνόδευτων, μη συνοδευόμενων ανηλίκων είναι και αυτό σημαντικό. Έχετε δικές σας δραστηριότητες που θα αναπτύξετε και θα αναλάβετε σίγουρα ε, σημαντικό ερώτημα αυτό. Τρίτος τομέας, η επανεγκατάσταση σε τρίτα κράτη αυτών των ανθρώπων. Πώς θα γίνει αυτό συγκεκριμένα και πώς αποκινούμε τα κράτη-μέλη που αφορούν αφορώνται άμεσα θα γίνει αυτή η δουλειά. Θα στείλετε συνεργάτες σας σε αυτές τις χώρες ή στις τρίτες χώρες ώστε να εξοικειωθούν με την κατάσταση επιτόπου και μία α το πω έτσι κάπως ε, διαφορετικού τόνου παρατήρηση. Αν έχουμε κάποιες ομάδες ή ε, κάποιες κατηγορίες που μας λένε πόσο τρομερά είναι τα πράγματα με τους ετούντες άσυλο και τους πάμπολους πρόσφυγες και μετανάστες δεν διαρωτάται κανείς τι συμβαίνει σε σχέση με την Ιταλία που αυξάνονται διαρκώς αυτοί οι αριθμοί και η Ιταλία προσπαθεί με κάθε τρόπο αυτούς να τους αποπέμψει. Ξέρω ότι είναι ίσως μειωτική αυτή η παρατήρηση, η τελευταία παρατήρηση, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό το πρόβλημα και να διατεθούν κονδύλια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Λάμπετ που είναι και συγγήτρια για το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, ευχαριστώ και τον ε, δόκτωρα Βίσερ. Μεγάλη είναι η χαρά μας που σας ξανασυνδαντούμε. Θα ήθελα και εγώ να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με τον προϋπολογισμό. Σε σχέση με αυτά που νομίζετε ότι δεν θα γίνουν ή με το τι θα έπρεπε να ε, γίνει πρώτο αν παραμείνει ο προϋπολογισμός ως έχει. Ε, ένα από τα ερωτήματα όταν ε, εξετάζαμε τον κανονισμό του ΕΑΣΟ και που δημιούργησε πολλά ερωτήματα γύρω από τις αιτήσει ασύλου και για τις πληροφορίες είναι το ζήτημα της διερμηνίας. Εμένα θα με ενδιέφερε πάρα πολύ να ξέρω ε, τι προσφέρεται από τα κράτη-μέλη ε, με ε, σκοπό να μπορούν να εξετάσουν τις αιτήσει αυτές καλύτερα, πιο αποτελεσματικά, ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί να εκφραστούν ευκολότερα. Το ζήτημα του συνοριακού ελέγχου δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά την ίδια την ΕΑΖΟ, αλλά θα ήθελα να σας ρωτήσω μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε ορισμένα πράγματα για τη σχέση της υπηρεσίας αυτής ε, με άλλους οργανισμούς που έχουν να κάνουν με μικτές μεταναστευτικές ροές, αν υπάρχουν τέτοιου είδους σχέσεις, αν αναπτύσσονται σιγά σιγά και αν είναι χρήσιμο να ε, δίνει μεγαλύτερη σημασία η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις μικτές ροές. Αν ακούσετε τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε, προσπαθούμε να περάσουμε από τον ε, έναν όρο στον άλλον και φυσικά ε, οι μικτές αυτές ροές μπορούν να συμπεριλάβουν πάρα πολλά πράγματα. Θα ήθελα λοιπόν να μας πείτε πώς μπορείτε να συνεργαστείτε με άλλα όργανα για να γεβηρωθούν αυτές οι διαφορές. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κλάες. Ευχαριστώ Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Πολύ Συμφωνώ ε, και εγώ με την ερώτηση του κυρίου Βάντερ Η κατάσταση στην, στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι ένα πρόβλημα το οποίο το σέρνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό και πρέπει να δράσουμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι ώστε ο ρόλος της Τουρκίας ως χώρα διαμετακόμισης και παράνομης μετανάστευσης να ενισχυθεί. Information report για τη χώρα προέλευσης. Θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η σκοπιμότητα Θα χρησιμοποιηθούν αυτές οι πληροφορίες για να αξιολογηθούν οι αιτήσει των πολιτικών ετούντων το άσυλο. Δεν βλέπω κανέναν άλλο να θέλει πάλι το λόγο, οπότε δίνω στον κύριο Βίσερ το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ κύριε ε, Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και τους ε, ευρωβουλευτές για τις ερωτήσεις τους. Θα προσπαθήσω να απαντήσω σε ερωτήσεις με τη σειρά που μου ετέθησαν θα προσπαθήσω να συνδυάσω τις ερωτήσεις για την Ελλάδα, γιατί υπήρξαν πολλές ερωτήσεις ε, που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αναφέρονταν στην Ελλάδα. Το ελληνικό ε, πρόγραμμα είναι ένα πολύ μεγάλο ε, εκτεταμένο πρόγραμμα που καλύπτει μία περίοδο δύο ετών περίπου Ενδεχομένω να, χρησιμο... να χρειαστεί και άλλο χρόνο, βέβαια γιατί είναι πάρα πολύ φιλόδοξο πρόγραμμα και αφορά τρία βασικά κεφάλαια σε σχέση με το άσυλο. Πρώτον, ε, τη δημιουργία ενό νέου οργανισμού ασύλου, μια νέα υπηρεσίας ασύλου. Δεύτερον, ε, μιας ε, ανεξάρτητης υπηρεσίας υποδοχής και επίσης με η αντιμετώπιση ε, του καταλόγου των ε, υποθέσεων που μένει ακόμη να εξεταστούν ε, στο άσυλο ε, γιατί υπάρχουν περίπου 15.000 αιτήσει οι οποίες δεν έχουν εξεταστεί ακόμη. Αν λοιπόν ε, το κατά πόσο είναι στεγανά τα σύνορα, όπως μας ρωτήσατε κύριε Φαντεν Κάμπ, είναι κάτι το οποίο δεν ε, μπορώ εγώ να σας απαντήσω. Μπορώ να επηρεάσω κάπως την κατάσταση στο πλαίσιο των μεικτών ροών, αλλά είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά βασικά τη Frontex. Η κυρία Λάμπερτ μας ε, με ρώτησε για τη σχέση μας ε, με τη, τους άλλους οργανισμούς. Η Frontex και εμείς ε, καταλήξαμε στο συμπέρασμα πολύ νωρίς ότι πρέπει να συνεργαστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο γιατί πράγματι πρόκειται για μικτές ροές και και εμείς και η Frontex έχουμε να αντιμετωπίσουμε τις μικτές αυτές ροές και όσο νωρίτερα φτάσουμε επί τόπου με παρακολούθηση, με ε, αναγνώριση, με τέτοιου είδους ε, ε, δράσεις, τόσο καλύτερα θα συνεργαστούμε. Και είναι πάρα πολύ σημαντική λοιπόν αυτή η συνεργασία και πράγματι κυρία Λάμπερτ αφορά τις μικτές ε, ροές ε, ε, και για μας και για τη Frontex. Οπότε ελπίζω να έχουμε μια διαδικασία ασύλου που θα οδηγεί και στην αποδοχή αλλά και στην απόρριψη αιτήσεων ασύλου συμπεριλαμβανομένης βέβαια της διαδικασίας επιστροφής των ανθρώπων αυτών. Τώρα, Ενάμιση με δύο μήνες έχουν περάσει ε, από τότε που πήγαμε στην Ελλάδα επί επιτόπου. Υπήρξαν κάποιες βελτιώσεις ε, όσον αφορά την ποιότητα των αποφάσεων. Η ύπατη αρμοστία του ΙΕ έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, βοήθησε πάρα πολύ. Υπήρξαν και πολλοί εμπειρογνώμονε από διάφορα κράτη-μέλη που ήταν παρόντες. Ε, Συγκεκριμένα αποτελέσματα, ναι, αλλά το να δημιουργεί κανείς ένα νέο οργανισμό μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ελκυστικός τρόπος για να δείξει σε κανέναν ότι αλλάζει η ποιότητα ή αλλάζουν οι αριθμοί. Πρέπει να υπάρξει πρώτα ένας σταθερός, ένας στέρεος οργανισμός για να μπορέσουν να υπάρξουν καλά αποτελέσματα και από τεχνικής απόψεως. Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι οι ελληνικές αρχές ε, δουλεύουν με πολύ επικοδομητικό και θετικό τρόπο προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν ξέρω τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γνωρίζω ότι είναι περίπλοκα τα πράγματα και από οικονομικής και από πολιτικής απόψεως, αλλά αυτή είναι ε, η απάντηση που μπορώ να σας δώσω και αυτά είναι τα στοιχεία που πρέπει να λάβω και υπόψη μου. Ε, για τον τομέα αυτών λοιπόν του ασύλου συγκεκριμένα είναι πάρα πολύ θετική και επικοδομητική η στάση των ελληνικών αρχών. Βέβαια παραμένει ακόμη πολύ δρόμος και δύο χρόνια είναι πολύς χρόνος. Όταν θα είναι το γραφείο μας πλήρως, ε, το πότε θα είναι ε, η υπηρεσία μας, συγγνώμη, πλήρως λειτουργική, Έχουμε περίπου 80 άτομα προσωπικό και ε, με τον ε, ε, προϋπολογισμό που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν νομίζω να τα καταφέρουμε την επόμενη εβδομάδα. Άλλωστε μπορεί να μειωθεί και ο προϋπολογισμός γιατί θα υπάρξει μηδενική αύξηση την επόμενη χρονιά. Οπότε πρέπει να δούμε, να περιμένουμε τουλάχιστον μέχρι το 2013 ελπίζοντας ότι τότε ο προϋπολογισμός ε, θα επανέλθει στα αρχικά του επίπεδα και θα μπορέσουμε και εμείς να προοδεύσουμε. Τώρα, το αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι βεβαίως ε, οι προτεραιότητες, τουλάχιστον ε, στη βασική δομή του οργανισμού, αλλά και επί του περιεχομένου αλλάζουν τα πράγματα, γιατί έτσι όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, του χρόνου που ελπίζουμε να επενδύσουμε στην εξωτερική διάσταση που είναι ένα σημαντικό τμήμα της ε, δουλειάς, ε, της δουλειάς μας. Ενδεχομένως οι προτεραιότητες ε, που θα ήθελα εγώ να έχω ως βασικές προτεραιότητες να μην μπορέσουν να βρίσκονται τόσο ψηλά στην ιεραρχία, στην ιεράρχησή μας. Θα ήθελα να πω επίσης ε, ότι Η βασική ευθύνη για συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις ε, επαφίεται πάντοτε στα κράτη-μέλη βάσει του κανονισμού αυτού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο. Ε, λαμβάνω βέβαια αιτήματα πολλά ήδη από τα κράτη-μέλη που δείχνουν τουλάχιστον το μεγάλο τους ενδιαφέρον για την υπηρεσία αυτή και ε, εκδηλώνουν και την υποστήριξή τους. Ε, ο κύριος Σαρκοζή δεν είναι μεταξύ αυτών ε, που μας έχει που, που μας, έχει απευθυνθεί, αλλά εν πάση περιπτώσει ποτέ δεν ξέρει κανείς. Όσον αφορά τον επιμερισμό του βάρους, αν δει κανείς την επανεγκατάσταση, όπως γνωρίζετε είναι κάτι το αρκετά ασαφές και μάλιστα αυτό έχει γίνει εσκεμένα στο πλαίσιο του κανονισμού γιατί πρόκειται για ζητήματα ιδιαίτερα πολιτικά Αναφέρεται λοιπόν στον ιδρυτικό κανονισμό ότι η ΕΑΣΟ θα διευκολύνει και θα συνεργάζεται ε, για την εφαρμογή κάθε απόφασης ε, αυτή τη στιγμή έχει ληφθεί. Βεβαίως η επίτροπο Μάλμστρομ και ε, η κυβέρνηση της Μάλτας ελπίζουμε να μα υποστηρίξουν όταν θα περάσουμε στην επόμενη φάση της επανεγκατάσταση. και πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να αφορά κυρίως τις αιτήσει που έχουν γίνει δεκτές, όχι γενικότερα τους ετούντες άσυλο, αλλά ε, τους, ε, τις αιτήσει άσυλο που είχαν ως αποτέλεσμα τη χορήγηση του ασύλου, τη χορήγηση την απόδοση του καθεστώτος του ασύλου σε, του, του ασύλου σε κάποιον συγκεκριμένο άνθρωπο, ε, όχι τις υπόλοιπες αιτήσει που, που είναι κρεμείς για τη συνεργασία τώρα στην Ελλάδα και με άλλους ε, εμπειρογνώμονες. Αυτό είναι πραγματικά το πολύ συναρπαστικό κομμάτι της συνεργασίας. Ε, οι εμπειρογνώμονες των κρατών μελών ε, Το να συνεργάζεται κανείς με εμπειρογνώμονε των κρατών μελών ε, είναι ε, ενδιαφέρον, ε, ακόμη και σε εθνικό επίπεδο μερικές φορές είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και συναρπαστικό. Ο δε συνδυασμό μεταξύ των εμπειρογνωμόνων ευρωπαϊκού επίπεδου και εθνικών εμπειρογνωμόνων είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον. τώρα η ενημέρωση απλώς δεν είναι επαρκής χρειάζεται μια διαχείριση συγκεκριμένη, ένα πρόγραμμα διαχείρισης ε, για να μπορέσει να καθοδηγηθεί η όλη διαδικασία. Αυτό είναι πραγματική ανάγκη και αυτό αποτελεί ένα καθήκον εμπειρογνώμονα και είναι κάτι το οποίο ε, πάντοτε, δεν έχουν πάντοτε όλοι οι αξιωματούχοι στο ε, εθνικό τους ενεργητικό, για να το πω έτσι ε, απάντησα νομίζω για τα ζητήματα της, ε, του προπολογισμού, τώρα για τη διερμηνία, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα. Η συνεισφορά της ΕΑΖΟ στο συγκεκριμένο θέμα, ε, κατά την άποψή μου, αφορά κυρίως την κατάρτιση, γιατί η κατάρτιση αποτελεί τη βάση αν έχουμε μια κοινή γλώσσα από απόψεως ε, πολιτικής, ε, μέσω της ε, κατάρτισης ενός κοινού προγράμματος ε, κατάρτισης ε, σε ολόκληρη την Ευρώπη, τότε εξασφαλίζουμε μία ελάχιστη κοινή γλώσσα τουλάχιστον. Όσον αφορά τώρα την οργάνωση των κοινών υπηρεσιών, όπως για παράδειγμα και ε, κοινή εκπαίδευση, αυτή συμπεριλαμβάνεται στις κοινές υπηρεσίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το πιλωτικό πρόγραμμα των, ε, αυτού του καταλόγου της ομάδας των διερμηνέων που θέλουμε να έχουμε για να δούμε καταρχάς ποια είναι τα υπέρ και τα κατά γιατί η διερμηνία είναι πάρα πολύ δαπανηρό μέσο και πρέπει να δούμε πώς θα μπορέσουμε να τη χρησιμοποιήσουμε με τον πλέον αποτελεσματικό τρόπο. Νομίζω ότι ήδη κάλυψα το θέμα της συνεργασίας με τη Frontex. Τώρα με τους υπόλοιπους οργανισμούς επίσης ε, θα θέλαμε να συνεργαστούμε, την Υπηρεσία Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, ενδεχομένως και με τη Europol αν χρειάζεται και όσον αφορά τις μικτές ροές, ε, την ε, σώματεμπορία, είναι ζητήματα για τα οποία συχνά συμφωνούμε και πρέπει να συνεργαστούμε και ελπίζω κάτι τέτοιο να συνεχιστεί και στο μέλλον. για το ρόλο της Τουρκίας τώρα. Κοιτάξτε, από τη φύση του είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Είναι μεγάλο και ευαίσθητο σύνορο. Είναι μια χώρα γειτονική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως η βασική, το βασικό ζήτημα εδώ είναι καθαρά ε, πολιτικό εξ όσων γνωρίζω, και στις ε, διμερείς σχέσεις μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, αλλά και μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Τουρκίας. Επομένως, ε, εμείς είμαστε μια απλή ευρωπαϊκή υπηρεσία και δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε τίποτε παραπάνω. Μπορεί να μην ε, απασχολήσει πάρα πολύ την υπηρεσία μας ε, στους επόμενους μήνες. Ενδεχομένως ασχοληθούμε με τη συνεργασία με τις γειτονικέ χώρες, ελπίζω και με την Τουρκία, ελπίζω να είναι μεγάλη προτεραιότητα για την ε, ε, ΕΑΖΟ, γιατί μπορούμε να είμαστε πολύ αποτελεσματικοί. Όσον αφορά τώρα τις εκθέσεις για το COI, δηλαδή για τις πληροφορίες της χώρας προέλευσης, αν καταφέρουμε να έχουμε μία αξιολόγηση της κατάστασης ε, στην χώρα προέλευσης, αυτό μπορεί να βοηθήσει τις ε, ε, αποφάσεις ήδη από την αρχή. Και έχω πολλές φορές μιλήσει με προσώπους της δικαστικής εξουσίας στην Ευρώπη και είναι πολύ ενθουσιασμένοι με αυτή την ιδέα του της κάποιας αξιολόγηση ε, της πληροφορίας που προέρχεται από την χώρα προέλευσης που δεν εξαντλείται μόνο σε μια έκθεση, <coughs> σε μια έκθεση αναχώρα εν πάση περιπτώσει. Οπότε... Είναι ένα πολύ, ένας πολύ φιλόδοξος στόχος. <coughs> Πρέπει όμως να δούμε και η κοινωνία των πολιτών και η ΜΚΟ, τα κράτη-μέλη, αλλά και το δικαστικό το δικαστικό ως παράμετρος. Ελπίζουν ότι θα έχουμε τέτοιες κοινέ αξιολογήσεις που θα τους βοηθήσουν να λαμβάνονται οι αποφάσεις, να δώσουν τις βάσεις για αποφάσεις στην Ευρώπη επί των ιδίων ε, βάσεων, είτε θα είναι στη Φινλανδία, Κύπρο, Ισπανία ή για οποιαδήποτε άλλη χώρα. Νομίζω αυτές ήταν οι ερωτήσεις και αυτές οι απαντήσεις μου. Ευχαριστώ. Thank you. Thank you. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση και τις επιπρόσθετες εξηγήσει. Αν δεν υπάρχει δεύτερη παρέμβαση, δευτερολογία από τα μέλη, αυτά είναι, ολοκληρώσαμε και σας ευχόμαστε και πάλι κάθε καλό και επιτυχία, κύριε Φίσερ, ώστε να καταφέρετε να συνεχίσετε με θετικό τρόπο το έργο που έχετε υποεξέλιξη. Συγγνώμη, δεν σας είχα προσέξει, δεν είσαστε στον κατάλογο, αλλά έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αλλά μου ήρθε ακριβώς ακούγοντας την ε, <coughs> απάντηση του, Προεδρε... του Προέδρου της ΕΑΣΟ. Ορισμένοι βουλευτές στην προηγούμενη θητεία εκτίμησαν και εν μέρη σε αυτήν εκτίμησαν ιδιαίτερα το γεγονός ότι οι μεταφράσεις θα πρέπει να γίνονται σε μία γλώσσα κατανοητή από τον ετούντα το άσυλο. Πέρα από, την ε, νομική, από το νομικό αντικείμενο που, για το οποίο δεν θα σας ρωτήσω τίποτα διότι συζητιέται ήδη πολύ το θέμα εδώ. Αλλά σε όλες αυτές τις περιπτώσεις που εσείς ε, διαπιστώνετε μέσα από την εμπειρία των 27 υπαλλήλων και άλλους που ζουν κοντά στους ετούντες στο άσυλο πιστεύετε ότι υπάρχουν προβλήματα έλλειψης κατανόησης των ετούντων ασύλου δηλαδή καταλαβαίνουν και συνεννοούνται καλά οι ετούντες στο άσυλο γίνεται κατανοητή η κατάσταση του ετούντος στο άσυλο. Έχετε τον λόγο να απαντήσετε κύριε Φύσερ. Σας ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Δεν ισχυρίζομαι σε αυτή τη χρονική στιγμή ούτε και στο μέλλον να έχω πραγματική γνώση για κάθε επιμέρους περίπτωση και για όλες τις περιπτώσεις αυτές. Θα μπορούσα όμως γενικότερα να πω κάτι ότι η διερμηνία έχει ζωτική σημασία στη διαδικασία χορηγήση ασύλου και θεμάτων ασύλου. Είναι το να έχουν το δικαίωμα οι άνθρωποι μια ευκαιρία να παρουσιάσουν το αίτημά τους με τον καλύτερο θετικό τρόπο και με υποστήριξη. Η διερμηνία λοιπόν είναι ένα ουσιοδέστατο στοιχείο σε όλα αυτά και υπό τα θεμελιώδη δικαιώματα και το πρίσμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και σε σχέση με μέρος της εργασίας του ε, οργάνου μας θα είναι να δώσουμε κίνητρα σε αυτό το τμήμα, σε αυτή την παράμετρο της διαδικασίας για τη διερμηνία χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα και χωρίς να υπάρχει και η επιθυμία να γίνουμε ένας παγκόσμιος, ένας πανευρωπαϊκός οργανισμός διερμηνίας δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό, ούτε θα ήταν και αποτελεσματικό σε σχέση με τα, τις δαπάνες. Λοιπόν, τονίζοντας και υπογραμμίζοντας πάντα την σπουδαιότητα, τη σημασία που έχει η διερμηνία, <clears throat> με την κοινή κατάρτιση που θα είναι τμήμα της δουλειάς για την κατάρτιση και τονίζοντας την ανάγκη να υπάρξει η διερμηνία και να εντάσσεται στο μέλλον σε αυτό το έργο, από πλευρά τη ΕΑΣΟ θα έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε, να θεσπίσουμε κατευθυντήριες γραμμές προς ανατολισμούς για τις υπηρεσίες για τα θέματα σύλλου πανευρωπαϊκά και θέματα σαν αυτό θα συναποτελούν τμήμα αυτών των διαδικασιών. Ευχαριστώ. Πρόεδρο σας, ευχαριστώ. Αυτό ήταν ένας, ε, μια δευτερολογία όσον αφορά την απάντηση σε δευτερολογία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε. Σας ευχαριστούμε κύριε Φίσερ. Ευχαριστούμε που ήρθατε και για την παρουσίαση του προγράμματος εργασίας 2011. Και προσβλέπουμε να σας ξαναδούμε και στο μέλλον ξανά. Γεια σας. Ευχαριστώ. then... Και θα έλεγα στη συνέχεια μπορούμε να προχωρήσουμε αμέσως στο επόμενο σημείο το οποίο είναι το σημείο υπαριθμών 18 στην ημερησία διάταξη και αφορά ένα θέμα που <clears throat> αναφέρεται στους ετούντες άσυλο και αυτό. Είναι η αναδιατύπωση του κανονισμού για ελάχιστους κανόνες και κανονισμούς για την υποδοχή των ετούντων άσυλο. Ο Αντώνιο Μασίπο, συνάδελφός μας ως εισηγητής και θα ακούσουμε από πλευράς του την παρουσίαση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξέρουμε ότι το 2008 είχε καταθέσει μια πρόταση για αναδιατύπωση της οδηγίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή της οδηγίας 2003 κάθετος 9 ε, για ελάχιστες προδιαγραφές για την υποδοχή ετούντων άσυλο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκλήρωσε την πρώτη, την πρώτη ανάγνωση τον Μάιο 2009 και για να προχωρήσουμε και να ανταποκριθούμε στην προθεσμία 2012 για την θέσπιση ενός κοινού συστήματος ε, για τους ετούντες άσυλο στην Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε μια αναδιατύπωση τροποποιημένη πρόταση κατά τη διάρκεια του Ιουνίου 2011. Ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κάνει μια σύντομη παρουσίαση αυτής της αναδιατύπωσης, τροποποίησης της πρότασης της Επιτροπής και αμέσως μετά θα ανοίξουμε τον γύρο παρεμβάσεων. Σημειώθηκε ότι από πλευράς Προεδρίας, που αφορά δηλαδή το Συμβούλιο, η Πολωνική Προεδρία θα φτάσει στις 4 ακριβώς, 16.00, 4 το απόγευμα. Όμως θα έλεγα για να μην κάνουμε κάποιο διάλειμμα ή καθυστερήσουμε και χωρίς να υπάρχει λόγος, ας παρακολουθήσουμε την παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μετά η Προεδρία θα μπορέσει να καλύψει το κενό σε σχέση με τη συζήτηση. Δεν θα είναι πρόβλημα αυτό. Εσείς έχετε τον λόγο κυρία, παρακαλώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Euh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Όπως το αναφέρατε αυτό το θέμα δεν είναι άγνωστο για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Μασίπη Ιντάλγο, τον εισηγητή, για όλη την δουλειά που έκανε επί της προτάσεως του 2008, όπως επίσης ευχαριστώ και το Κοινοβούλιο για την υποστήριξή του το Μάιο του 2008 για την πρόταση αυτή. Όπως γνωρίζετε, οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο δεν έτυχαν της ίδιας επιτυχίας το Συμβούλιο δεν κατάφερε να καταλήξει σε μια κοινή θέση. Γι' αυτό λοιπόν η Κομισιόν αποφάσισε να αναλάβει τις πολιτικές της ευθύνες και να ασκήσει το δικαίωμα πρωτοβουλίας για να μπορέσει να δώσει μια νέα όθηση στις εργασίες με μια τροποποιημένη πρόταση της 1ης Ιουνίου πρέπει να διπλασιάσουμε την προσπάθειά μας για να καταφέρουμε να προσεγγίσουμε το στόχο του 2012 και πιστεύουμε ότι είναι απόλυτα δυνατόν να ορίσουμε ένα κοινό καθεστώς ασύλου στην Ευρώπη που να είναι και δίκαιο και αποτελεσματικό για τους ετούντες το άσυλο αλλά και για τις αρχές των κρατών μελών. Η τροποποιημένη πρόταση της 1ης Ιουνίου λαμβάνει υπόψη της στη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2009 και των συζητήσεων στο Συμβούλιο όπως επίσης και των επιπλέον διαβουλεύσεων που, στις οποίες προχώρησε η Κομισιόν τους τελευταίους μήνες. Οι δύο μεγάλοι στόχοι αυτής της πρότασης ε, ε, είναι αφενός να διατηρήσουμε την προστιθέμενη αξία της εναρμόνισης, δηλαδή να προχωρήσει περισσότερο από την τωρινή οδηγία του 2003 και επίσης να καλύψει και τα ελλείμματα τα οποία είχαμε διαπιστώσει κατά την αξιολόγηση της εφαρμογής. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα υψηλότερο επίπεδο συγκρισιμότητας και περισσότερες πρόοδους στο σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η τροποποιημένη πρόταση λαμβάνει υπόψη το θέμα της κράτησης και τις ανάγκες των, των πιο αδύναμων ατόμων. Θέλουμε να διευκολύνουμε ορισμένους κανόνες να γίνουν πιο ελαστικοί για, για να μπορέσουν να εφαρμοστούν σε επίπεδο εθνικού δικαίου. Αυτό ήταν και ένα πρόβλημα που είχαμε αντιμετωπίσει στο Συμβούλιο. Υπάρχουν διαφορές στις πρακτικές των κρατών μελών και θέλουμε να έχουμε την εποπτεία της οδηγίας από την Κομισιόν. Η πρόταση έχει κανόνες που επιτρέπουν στα κράτη-μέλη που υπόκεινται ιδιαίτερες μεταναστευτικές ροές να έχουν στη διάθεσή τους τα απαραίτητα μέσα για να μπορούν να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά και πάντα στο ίδιο πλαίσιο εμείς λάβαμε υπόψη μας περισσότερο τα οικονομικά και δικητικά άχθη που προκύπτουν από την πρόταση της Κομισιόν. Πιο συγκεκριμένα θα ήθελα να σας αναφέρω τέσσερις μεγάλες κατηγορίες τροπολογιών στη θέση της 1ης Ιουνίου. Πρώτη μεγάλη κατηγορία αφορά στους κανόνες εκείνους οι οποίοι είναι ήδη καθαροί, διευκρινισμένοι και παραμένουν ίδιοι. Η Κομισιόν ανησυχεί για την συχνή κράτηση των ετούντων ασύλου και η Λίμπε επίσης ανέφερε τις ανησυχίες της σχετικά συχνά και αυτό μετά από πολλές επισκέψεις στα διάφορα κέντρα κράτησης ανά την Ένωση. Πρέπει να διατηρήσουμε σαφείς και εναρμονισμένους κανόνες για την κράτηση ώστε να εφαρμόζεται πιο αρμονικά και να είναι και ένα μέτρο τελευταίες χάτης ανάγκης. Αυτή η πρόταση διατηρεί τον όρο που λέει ότι η κράτηση επιτρέπεται μόνο όταν έχουμε ορισμένους ε, λόγους ε, που καλύπτονται από την οδηγία ισχύει η αρχή της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας που πρέπει να, που πρέπει να αποδειχθούν και χρειάζεται γρήγορη πρόσβαση στη δικαιοσύνη και απαραίτητη δικαστική βοήθεια. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να είναι σύμβατες με τη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων αλλά και την πρόσφατη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα. Ταυτόχρονα η τροποποιημένη πρόταση είναι πιο ευέλικτη όσον αφορά στην κράτηση που εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές και όπου είναι δύσκολο στην πράξη να προσφέρουμε όλη την γκάμα των ε, εγγύσεων που προσφέρονται και αυτό ισχύει για, ε, για τα διαμετακομιστικά κέντρα και για τα συνοριακά φυλάκια. Θέλουμε να έχουμε αξιοπρεπείς διαδικασίες για τους ε, ετούντες στο άσυλο η πρόταση λέει ότι θα πρέπει να εφαρμοστούν εθνικά μέτρα για την γρήγορη διαπίστωση των αναγκών υποδοχής των ε, ευάλωτων ατόμων και να παρακολουθείται η κατάστασή τους στη συνέχεια. Οι κανόνες για τη διαπίστωση ε, εκφράζονται με απλούστερο τρόπο δεν ορίζουν αυτόματα τη λήψη διοικητικών μέτρων και μπορούν κάλλιστα να ενταχθούν στον κατάλογο των, εθνικών, ε, των υπαρχών των εθνικών νομοθεσιών. Αυτό μας το ζήτησαν πολλά κράτη-μέλη στο Συμβούλιο. Ο ορισμός των ανθρώπων με ειδικέ ανάγκες και αυτός διευκρινίστηκε. Υπογραμμίζω ότι λαμβάνοντας υπόψη το ψήφισμα του Μαΐου του 2009 δεχόμαστε την ισοτιμία στην πρόσβαση των δικαιωμάτων ε, στην υγεία. Είχαμε διαπιστώσει παλιότερα ότι υπήρχε ένα πρόβλημα με την ηλική βοήθεια που δίνουν τα κράτη-μέλη στους ετούντες στο άσυλο και οι διατάξεις που έχουμε σήμερα είναι αρκετά ασαφείς και δημιουργούν διαφορετικές πρακτικές. Θέλαμε κατά συνέπεια να, διατηρήσουμε, να θέσουμε έναν ορισμό του τι είναι κατάλληλος τρόπος ζωής για να μπορείτε να, να, δίνετε και η απαραίτητη αποζημίωση. Για την θέση τώρα του Κοινοβουλίου και για τη θέση του Συμβουλίου η τροποποιημένη πρόταση δεν αποτελεί ένα ενιαίο σημείο αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάθε κράτος μέλος είναι αυτό που πρέπει να ορίζει συγκεκριμένα κριτήρια σε εθνικό επίπεδο. Αυτά τα κριτήρια όμως πρέπει να είναι μετρήσιμα και να επιτρέπουν την παρακολούθηση της βοήθειας που παρέχεται στους ετούντες μια διαφοροποιημένη μεταχείριση των ετούντων άσυλο έναντι των εθνικών υπηκόων είναι δυνατή, φτάνει να είναι και σωστά και διαφανώς ε, δικαιολογημένη. Η άλλη ομάδα τροποποίησεων στην τροποποιημένη πρόταση θέλει να ευνοήσει μια μεγαλύτερη αυτονομία των ετούντων το άσυλο. Αυτό αυτό σημαίνει ότι η Κομισιόν συνεχίζει να θεωρεί ότι η ανεργία που επιβάλλεται στους ε, ετούντες στο άσυλο λόγω των κοινωνικών επιδομάτων και των αποζημιώσεων επιβαρύνει αδίκως τα κράτη-μέλη. Αυτή η επιβεβλημένη ανεργία μειώνει τα φορολογικά έσοδα διότι ευνοεί τη μαύρη εργασία θεωρήσαμε ότι η πρόσβαση στην απασχόληση είναι καλό και για τον ετούντα το άσυλο και για το κράτος υποδοχής. Εμείς κρατάμε αυτή την προθεσμία των έξι μηνών για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Σύμφωνα και με την πρόταση του Κοινοβουλίου επιτρέπουμε μία παράταση του ενός έτους για τους μη συνεργαζόμενους ε, ετούντες ή αν έχουμε πολλούς ετούντες στο άσυλο μαζί. Και αυτό είναι και συμβατό με την τροποποιημένη πρόταση που εγκρίθηκε την 1η Ιουνίου για την οδηγία διαδικασίας ε, για το άσυλο που θα το δούμε όμως μια άλλη φορά η τελευταία ομάδα τροπολογιών σημαίνει, ε, ε, στοχεύει στην απλούστευση απλούστευση που απέτησαν τα κράτη-μέλη όταν, από τη στιγμή που είχαμε και την πρώτη έκδοση της οδηγίας. Η πρόταση δίνει ένα μεγαλύτερο περιθώριο χειρισμών στην εφαρμογή και λαμβάνει υπόψη, όπως είχα πει στην αρχή, τις διοικητικές υποχρεώσεις και τις οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν για τα κράτη-μέλη που δέχονται ιδιαίτερες μεταναστευτικές πιέσεις έχουμε καλύτερες, καλύτερους νομικούς ορισμούς για την υποδοχή ε, και πιο ευέλικτους ε, κανόνες ε, για τις εθνικές πρακτικές. Συμπερασματικά κύριε Πρόεδρε, η πρόταση θα πρέπει να εξεταστεί παράλληλα με την ε, οδηγία για τη διαδικασία του ασύλου και ε, με υπό το όμα του Βουβλίνου. Αυτή η τροποποιημένη πρόταση οδηγεί σε μια ισορροπία μεταξύ της αποτελεσματικότητας του συστήματος ασύλου και της μεγαλύτερης προστασίας για τους ετούντες το άσυλο έτσι όπως ε, απαιτείται από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Τελειώνοντας θέλω να διασφαλίσω τον εισηγητή αλλά και τα μέλη της Επιτροπής σας για την, εργασία της, ε, για την προθυμία της Κομισιόν να συνεργαστεί μαζί σας και θα διευκολύνουμε ε, μεσολαβώντας για τη συμφωνία των δύο συνομοθετών τον επόμενο μήνα. Ευχαριστώ κύριε Αγγέλ, θα ακούσουμε τον κύριο Μασίπ, τον εισηγητή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για μένα ως εισηγητή, ήδη στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία για την οδηγία, για την πρόταση που τροποποιήθηκε και τροποποιήθηκε τώρα, εκείνο που με ενδιαφέρει είναι σε σχέση με τους ε, συναδέλφους της Επιτροπής και την ίδια την Επιτροπή και το Συμβούλιο τουλάχιστον σε σχέση με την εκπροσώπηση από πλευρά του ε, επιφανούς φίλου. Θα πρέπει να εντάξουμε όλα αυτά τα θέματα νομικά στην ιστορία των όσων συνέβησαν στο παρελθόν. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία είχαμε ένα μεγάλο επίτροπο, τον κύριο Μπαρνιέ, που έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια. Συγγνώμη, συγγνώμη ο Μπαρό, ο κύριος Μπαρό, ο επίτροπος. Ε, λοιπόν, εντάξει. Ο κύριος Μπαρό, λοιπόν, ενεπλάκη, είχε εμπλακεί πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό σε αυτό το κείμενο, σε αυτό το κείμενο που τώρα τροποποιήθηκε. Μέχρι εκείνη του σημείου όπου σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή εγώ το είχα, το έβλεπα, το είχα χάσει, το θεωρούσα όχι σε, σε σχέση με την Επιτροπή Λίμπε, γιατί η Επιτροπή Λίμπε είχε πάντα πολύ μεγάλη ευαισθησία για τέτοιου είδου θέματα. Όμω το υπόλοιπο κοινοβούλιο βρήκαμε και είδαμε ότι βρεθήκαμε σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη για να προχωρήσει αυτή η έκθεση. Ο Μπαρό, ο Ζακ Μπαρό λοιπόν είναι εκείνος που είχε εμπλακεί ιδιαίτερα στην ίδια την Ολομέλεια βοηθώντας με στην υπεράσπιση που χρειάστηκε να κάνω στην Ολομέλεια για αυτά τα θέματα και την τελευταία στιγμή προχωρήσαμε και μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία. Τώρα, συνειδητοποιώντας με τις ε, ε, ε επιλογές αυτές ήξερα ότι θα μειωνόταν, θα είχε κάποια συρρήκνωση και ότι θα συνέβαινε αυτό το οποίο συνέβη τελικά. Τώρα, εν πάση περιπτώσει, είχαμε την τεράστια τύχη εκείνη που είμαστε υπέρμαχοι του να, να υπερασπιστούμε το άσυλο σε σχέση με τις προτάσεις στα κείμενα. Είμαστε όλοι υπέρμαχοι του ότι θα έπρεπε με μεγάλη δραστηριοποίηση και ενεργοποίηση και για την την παρουσία της Σεσίλια Μάρμστρομ ενώπιον της Επιτροπής ε, της Επιτροπής ε, που είχε επιφορτιστεί για την αναδιατύπωση αυτού του κειμένου. Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών εργαστήκαμε και εγώ είδα αυτή τη γυναίκα. Την είδα να εμπλέκεται σε βάθος με όλη της την ψυχή στο να αναζητήσει, να αναζητηθεί μια λύση με τα κράτη-μέλη στο Συμβούλιο θετική στα κράτη που είχαν τα εμπόδια και έθεταν τα εμπόδια που τώρα γνωρίζουμε όλοι ποια είναι. Αισθάνομαι λοιπόν υποχρεωτικά και πρέπει να τα πω αυτά, διότι ενώ πρέπει να προχωρήσουμε για αυτό το θέμα, πρέπει να είμαστε και πρακτικοί και να είμαστε ρεαλιστέ. Προφανώ θα συνεχίσω να συνεργάζομαι με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με τη Σεσίλια Μάρμστρον και φυσικά και με το Συμβούλιο. Και θα έχουμε και μια συνέντευξη που θα έχω με τον ε, εκπρόσωπο της Πολωνίας για αυτά τα θέματα, σίγουρα. Θα δούμε λοιπόν να καταφέρουμε κάτι αυτούς τους έξι μήνες. Θα τα καταφέρουμε, αλλά από την άλλη πλευρά είναι σε αυτή τη διαδικαστική στιγμή σαφές ότι υπάρχουν ζητήματα τα οποία βρίσκονται πολύ πιο πέρα από αυτά που ο εισηγητής θα έπρεπε να δεχτεί και μπορούσε να δεχτεί. Για παράδειγμα, αυτό το οποίο αναφέρθηκε από την εκπρόσωπο της Επιτροπής μόλις τώρα, στον συνεκτικό λόγο που μας ε, ε, παρουσίασε. Τι μας είπε. Μας είπε ότι η δουλειά που γίνεται σε σχέση με τους μετανάστες, η πρόσβαση στην εργασία, όχι μόνο θα είχαμε περιορισμό έξι μηνών, που προηγούμενα είχε τεθεί, αλλά προβλέπονται και άλλοι έξι μήνες επιπρόσθετοι ώστε, ας το πω έτσι, με έναν τρόπο υπερβολικά ελαστικό να μπορούν να μην έχουν πρόσβαση σε εργασία. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι απαράδεκτο. Τουλάχιστον σε αυτή τη διαδικαστική για μένα από πλευρά μου. Παρότι και εγώ είμαι ανοιχτό και πρόθυμο για λύσει που πρέπει να επιληθεί αυτό το πρόβλημα, να δούμε πώ θα επιληθεί. Το δεύτερο θέμα είναι οι όροι και προποθέσει για την αξιοπρέπεια, για τις κοινωνικές προϋποθέσεις και όρους που θα αντιμετωπίζονται οι αιτούντες άσυλο και που με την πλειοψηφία σε σχέση με την προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία θα μπορούσαν να, ίσως να μην έχουν αυτού του είδους την κάλυψη. Όπως ε, αναφέρθηκε και από την, Επίτροπο της, α, την της Επιτροπής, πρέπει να είμαστε σε γρήγορση. Τι θα συμβαίνει αυτό σε τέλος τέλος η διαφοροποίηση αυτή σε σχέση με τους ετούντες άσυλο. Και το τρίτο θέμα το οποίο θα έπρεπε να μας απασχολήσει κάπως περισσότερο και να εκφράσουμε τα μελήματά μας στην επανένωση οικογενειών και εδώ θα πρέπει να αναφερθώ στην έκθεση Λάμπερ που εγκρίθηκε χθε και που πρέπει να καταλήξει σε σχέση με την διατύπωση που θα πετύχουμε όλοι μας να μας επηρεάσει και σε αυτό. Λοιπόν, συνοψίζω και θέλω να πω, είμαστε πρόθυμοι φυσικά ανοιχτοί να καταλήξουμε σε προτάσεις, με προτάσεις σε ένα νέο κείμενο και με την, τον εκπρόσωπο της Πολωνίας, Πολωνικής Προεδρίας, αλλά με τις ιδιομορφίες αυτές που ανέφερα πιο πριν, με αυτά τα στοιχεία. Και τις ε, προσπάθειες της Επιτρόπου με θετικό τρόπο τις βλέπουμε και της Επιτροπής γενικά και μας ικανοποιεί ιδιαίτερα ότι όπως ακούσαμε από τον εκπρόσωπο της ΑΣΟ ε, πριν πρέπει το κοινοτικό εκτιμένο να ληφθεί υπόψη και το θέμα της διερμηνίας είναι τεράστια σημασία για μας. Ευχαριστώ. Αυτά ήθελα να πω. Σας ευχαριστώ κύριε Μασίπη Σίγητα και τώρα καλωσορίζουμε εσάς ε, τον εκπρόσωπο της Πολωνικής Προεδρίας που έχει την Προεδρία στο Συμβούλιο φτάσατε στην Επιτροπή μας, είσαστε καλοδεχούμενοι. Συζητούμε αυτό το θέμα, την αναδιατύπωση της ε, πρότασης για τις ελάχιστες προδιαγραφές για την υποδοχή ετούντων άσυλο. Αναμένουμε για να ακούσουμε από πλευρά σας ε, ποιες είναι οι θέσεις της Προεδρίας του Συμβουλίου. Είσαστε έτοιμοι να παρέμβετε. Παρακαλώ. Um, uh, uh, Ευχαριστώ πολύ και καλησπέρα σε όλους. Περιμένουμε την αναθεωρημένη εκδοχή του κειμένου μέχρι τα τέλη του... Περιμέναμε μέχρι τα τέλη του Ιουνίου. αλλά θέλουμε οι διαπραγματεύσεις ε, να διεξαχθούν το συντομότερο δυνατόν και όσο το δυνατόν ε, πιο αποτελεσματικά. Θέλουμε σε επίπεδο εμπειρογνωμόνων να γίνει η πρώτη ανάγνωση στο Συμβούλιο κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Αυτό έχει ήδη γίνει και επί τη βάση της συζήτησεως ε, να αρχίσουμε να συζητούμε τις συμβιβαστικές ε, προτάσεις που μπορούν να υποβληθούν στα κράτη-μέλη. Αυτό θα κάνουμε κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών και θα παρουσιαστούν ε, στο, στους εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου το Σεπτέμβριο. Αυτό είναι το πρώτο μας πρόγραμμα και θα δούμε τι πρόοδο μπορούμε να σημειώσουμε με βάση αυτά. Όσον αφορά τώρα την ουσία της συζήτησης θεωρούμε ότι μέχρι στιγμής ε, υπήρξε επικοδομητική στο πλαίσιο του Συμβουλίου και ότι βέβαια πρέπει να γίνει ακόμη πολλή δουλειά σε σχέση με τα εκκρεμή ζητήματα, τα πιο δύσκολα ζητήματα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει δυνατότητα περαιτέρω εργασιών και ελπίζουμε ότι κατά τη διάρκεια του Σεπτέμβρη και του Οκτώβρη θα, ε, θα υπάρξει πρόοδος. Ευχαριστώ. Και εγώ ευχαριστώ λέει ο πρόεδρος. Ο κύριος Παπα-Νικολάου θέλει να πάρει το λόγο. Thank you, Allow Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω στα ελληνικά. Θέλω να ευχαριστήσω την Επιτροπή για την εισήγησή της, να ευχαριστήσω και τον εισηγητή μας και να προσθέσω και εγώ από την πλευρά της, δική, της δικής μας πολιτικής ομάδας, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, κάποιες γενικές κατευθύνσεις το πρώτο είναι ότι όλοι συμφωνούμε ότι θέλουμε να προχωρήσουμε με το πακέτο ασύλου και θέλουμε να το κάνουμε και γρήγορα. Και αυτό όχι μόνο γιατί έχουμε συμφωνήσει σε ένα πολιτικό επίπεδο ότι το 2012 πρέπει να έχουμε ολοκληρώσει, αλλά και γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι η περίοδος αυτή είναι ιδιαίτερος πιεστική και κρίσιμη σε σχέση με τους ε, πολλούς συνανθρώπους μας δυστυχείς και ταλαιπωρημένους που καταφθάνουν στην Ευρώπη από τις γύρω περιοχές και με ε, όσα συμβαίνουν ε, και τις αναταραχές και στη Βόρεια Αφρική και στη Συρία και στις γειτονικέ χώρες. Ακριβώς για αυτούς τους λόγους είμαστε διατεθειμένοι να ε, καταθέσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να ολοκληρώσουμε μελετούμε προσεκτικά τι συνέβη το προηγούμενο διάστημα. Εγώ δεν ήμουν εδώ στην προηγούμενη Βουλή, ε, στην προηγούμενη θητεία. Ε, προσπαθώ όσο μπορώ να μελετήσω όμως τι συνέβη τότε, ποιε ήταν οι δυσκολίες, πού ακριβώς κολλήσαμε στο Συμβούλιο και πώς μπορούμε κι εμείς επικοδομητικά να συνεισφέρουμε προς την κατεύθυνση της συνένεσης και της συμφωνίας στις βασικές κατευθύνσεις. Ωστόσο, οφείλουμε όμως παράλληλα να έχουμε υπόψη μας κείμενα που μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί από το Κοινοβούλιο μας, τοποθετήσεις συγκεκριμένες που έχουν υπάρξει στο προηγούμενο διάστημα και ε, ο καθένας από εμάς ξεκινάει με κάποιες αφετηρίες και προφανώς στο τέλος όλοι θα επιδιώξουμε τη σύνθεση. Ε, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι πρέπει να προστατέψουμε αυτούς τους ανθρώπους. Ότι πρέπει να έχουν τα δικαιώματα που τους αρμόζουν. Ότι οφείλουμε να δούμε, ειδικά σε κάποια κράτη-μέλη που δεν είναι επαρκής η προστασία, να είναι εκείνη που πρέπει η προστασία. Ε, στα πλαίσια όμως των σκέψεων που κάνουμε και των αποφάσεων που θέλουμε να λάβουμε, οφείλουμε να προσπαθούμε να έχουμε μία συνοχή. Και τι εννοώ. Δεν μπορούμε άλλα να πούμε σε αυτή την ε, σε αυτή την έκθεση και άλλα να λέμε στην έκθεση για παράδειγμα της κυρίας Γκυγιόμ ή άλλα να λέμε σε αυτή την έκθεση και στην έκθεση για τους εποχικούς εργαζόμενους να έχουμε τώρα τροπολογία ότι εκείνοι που αναμένουν την, ε, την ε, απάντηση για το αίτημά τους για το άσυλο θα μπορούν στο μεσοδιάστημα με βάση τροπολογία θα κρυθεί αυτό αν θα εγκριθεί στην πορεία θα μπορούν να είναι εποχικοί εργαζόμενοι. Παράδειγμα, αυτό δημιουργεί ε, μία, αν μου επιτρέπετε, ε, έλλειψη συνοχής και νομίζω ότι δεν μας διευκολύνει στο να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κοινούς τόπους και κοινά συμπεράσματα. Αυτό που τέλος θέλω να πω, έχω πολλές παρατηρήσεις για τα επιμέρους ζητήματα, νομίζω δεν είναι τις παρούσε επειδή είναι η πρώτη εισήγηση. Αυτό που θέλω να πω κλείνοντας είναι ότι πέραν του, του τι θέλουμε να επιτύχουμε πρέπει να δούμε και τι μπορούμε να υλοποιήσουμε. Υπάρχουν βεβαίως ε, οι διαπιστώσεις που έχουν γίνει, υπάρχουν παραδείγματα καλά από κάποιες πρακτικές εθνικές, υπάρχουν κακά παραδείγματα ο πρώτος που αποδέχεται κακά παραδείγματα είμαι εγώ που προέρχομαι από την Ελλάδα και ξέρετε και τις καταδικαστικές αποφάσεις που υπάρχουν. Βεβαίως να κάνω εδώ μια παρένθεση και να πω ότι δεν είναι δυνατό να κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια να προχωρήσουμε και να παραμένουμε στάσιμοι και να παραμένουμε σε αδιέξοδο ό,τι αφορά το Δουβλίνο 2. Εν πάση περιπτώσει, ε, Κλείνοντα, θέλω να πω αυτό. Στα πλαίσια λοιπόν των πραγματικών συνθήκων και των αναγκών που υπάρχουν και της προσδοκίας όλων μας να προστατέψουμε με τους καλύτερους δυνατούς όρους τους συνανθρώπους μας που φτάνουν στην Ευρώπη έχοντας ανάγκες και προβλήματα, ε, με αυτούς τους όρους θα καταθέσουμε και εμείς κάθε δυνατή προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. Again. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Λάμπερτ και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για μια πάρα πολύ σαφή επεξήγηση της αναδιατύπωσης, της αναδιατύπωσης ώστε να δούμε ποιες είναι οι αλλαγές που έχουν γίνει. Αλλά όπως είπαν και πολλοί συνάδελφοι, στο... εδώ στο Κοινοβούλιο πρέπει να δούμε τη θέση που έχουμε ήδη ενώπιόν μας και να δούμε τις νέες προτάσεις για να δούμε ποια θα είναι και η προσέγγισή μας, πώς θα τοποθετηθούμε επί αυτών. Ε, θα... Σε σχέση λοιπόν με τις ιδέες που μπορούμε να έχουμε, καταρχάς πρέπει να είμαστε συνεκτικοί, να υπάρχει μια συνοχή και με τις διαδικασίες αλλά και με το Δουβλίνο. Για μας ως Επιτροπή αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δούμε πώς θα το κάνουμε αυτό να υπάρχει αυτή η συνεκτική προσέγγιση, όπως ήδη υπόθηκε από συναδέλφους επίσης, αναφέρθηκε τουλάχιστον ε, το θέμα του ορισμού της οικογένειας, που είναι κάτι το οποίο, στο οποίο δεν ε, πήραμε ακριβώς αυτό που θέλαμε από το Συμβούλιο, αλλά υπήρξε κάποια πρόοδο σε σχέση με τα γλωσσικά θέματα και με σε μερικούς άλλους τομείς ε, που εμφανίζονται στην πρόταση αυτή. Έχουμε τώρα πολύ εκτενείς αξιολογήσεις ε, του πώς λειτουργεί η οδηγία αυτή στα διάφορα κράτη-μέλη, με τα διάφορα προγράμματα. Έχουμε πολλά προγράμματα που μας επιτρέπουν να αξιολογήσουμε την κατάσταση σε σχέση με την πρώτη φορά που εξετάσαμε την κατάσταση αυτή, την πρώτη αναδιατύπωση δηλαδή, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία. Επίσης, θα ήθελα να πω ότι χαίρομαι που το Συμβούλιο έχει αυτή την προσέγγιση ότι θα τα καταφέρουμε ως προς αυτό που είναι πραγματικά μια πολύ ε, ευχάριστη, ευπρόσδεκτη προσέγγιση σε σχέση με άλλου είδους προσεγγίσεις που είχαμε ακούσει στο παρελθόν. Τώρα πρέπει να δούμε κατά πόσο ορίζουμε την πρόοδο με τον ίδιο τρόπο, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ θα ήθελα κάποια καθοδήγηση σε σχέση με τη διαδικασία που θα ακολουθήσουμε ως κοινοβούλιο κατά την εξέταση του θέματος αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Σίπελ. Ναι, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα καταρχήν <laughs> Δύο λόγια να πω για αυτά τα οποία προανέφερε ο κ. Παπα-Νικολάου για τη συνεκτικότητα και συνάφεια διαφορετικών μέτρων. Δύο λόγια θα ήθελα να πω σε σχέση με το θέμα των δυνατοτήτων σε τον άσυλο. Και θα έλεγα θα έπρεπε κυρίως μία συνεκτικότητα να υπάρχει εδώ όποιος ε, βρίσκεται νόμιμα στα κράτη-μέλη μας πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και να εργαστεί. Και αν έχει αυτό το δικαίωμα θα πρέπει η αρχή, η απλή αρχή, ίδιος μισθός για την ίδια δουλειά σε κάθε τόπο να ισχύει, άσχετα για την προέλευση και την ε, ε, ε και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ακούσαμε αρχικά κάποια συγκεκριμένα στοιχεία που αφορούν αυτό το νέο κείμενο το οποίο τροποποιήθηκε τώρα προς ποια κατεύθυνση κινούμαστε και με ικανοποιεί ότι αναμένει και μάλιστα αδειμονεί να ασχοληθεί η νέα Προεδρία με αυτό το κείμενο. Δεν άκουσα όμως προς ποια κατεύθυνση στοχεύει η νέα Προεδρία να κατευθυνθεί σε αυτό το κείμενο. Θα ήμουν ευγνώμων να μας έδινε το ένα ή άλλο στοιχείο πιο συγκεκριμένα η Προεδρία. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, επιτρέψτε μου και εμένα αφού και με τις άλλες οδηγίες ασχολήθηκα, να ασχοληθώ και με αυτή την οδηγία για τους όρους ε, υποδοχής ε, για τους ε, μετανάστες και επιτρέψτε μου για τη συνεκτικότητα με τις προηγούμενες αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου όπως ανέφερε ο εισηγητής ένα τμήμα έγινε δεκτό, ένα άλλο τμήμα όμως όχι το τμήμα το οποίο δεν εντάχθηκε ήταν παράδειγμα ότι δεν προβλέπεται ισότιμη θέση για τις κοινωνικές παροχές. Γιατί για κάποιες χώρες πάει πολύ μακριά αυτό και θα ήταν δύσκολο να υλοποιηθεί και θα δημιουργούσε απαιτήσει οικονομικές. Αλλά συμφωνήσαμε τουλάχιστον ότι από πλευράς Ευρωκοινοβουλίου θα πρέπει να υπάρχει μια αξιοπρεπής ε, ε, κάλυψη των αναγκών των ε, ετούντων άσυλο. Και για εκείνους που καταλήγουν σε εμά και ζητούν ζητούν άσυλο θα πρέπει με αξιοπρέπεια να αντιμετωπίζονται και να έχουν όρους διαβίωσης αξιοπρεπής. Η κυρία Λάμπερτ έθιξε την έννοια της οικογένειας μέσα σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να είμαστε συνεκτικοί πραγματικά στην οδηγία για τους όρους και προϋποθέσεις συμφωνήσαμε για τη θέση και στο τέλος τέλος που το Συμβούλιο ήταν ε, πρόθυμο να υιοθετήσει. Σε διαφορετικές οδηγίες δεν πρέπει να έχουμε διαφορετικούς ορισμούς για τις οικογένειες, διότι είναι δύσκολο να έχουμε έναν ορισμό σε μια οδηγία για την οικογένεια, άλλον ορισμό για μια άλλη οδηγία για την οικογένεια. Υπάρχει κάτι που με εκπλήσει το ότι βρίσκεται ακόμα αυτό εκεί ο τομέας δηλαδή της δωρεάν νομικής συνδρομής. Είχαμε μια άλλη ε, πορεία και διακομματικά, διακοινοβουλευτικά ε, συμφωνήσει ώστε να υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών οδηγιών για την δωρεάν συνδρομή. Διότι πρακτικές λύσεις πρέπει να υπάρχουν, εφικτές και πρακτικές λύσεις και όχι να περιμένουμε μέχρι το 2014 να μην γίνεται τίποτα επειδή δεν μπορούν να συνδιαλλαγούν μεταξύ τους οι διάφορες ομάδες. Το πακέτο αυτό πρέπει σε πλήρες πλαίσιο με πάγιες ε, συνθήκες ε, και όρους και προϋποθέσεις να λειτουργήσει ώστε να αξίζει τον τίτλο δίκαιο περί ασύλου, δίκαιο για τους ετούντες άσυλο. Αυτό το οποίο βρίσκω ότι είναι προβληματικό είναι επανειλημμένα το θέμα του ασύλου να συγχέεται με θέματα μετανάστευσης, γενικά με τη μετανάστευση. Το ένα είναι ανθρωπιστικό δίκαιο και το άλλο είναι θέμα μετανάστευσης, δηλαδή πώς θα αντιμετωπίσουμε τα θέματα αγορών εργασίας και των αναγκών που έχουμε για εργατικό δυναμικό. Πρέπει να υπάρχει διαφοροποίηση. Να μην συγχαίουμε τα πράγματα και τα ρίχνουμε όλα σε ένα καζάνι, σε μια οδηγία. Να διαφοροποιούμε πολύ προσεκτικά το ένα από το άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω για τις νέες προτάσεις που μας έχει παρουσιάσει και παρόλο που χρειάζεται να μελετηθούν αυτές σε λεπτομέρεια, παίρνω θάρρος από την προθυμία της ε, νέας ε, πολωνικής προεδρίας να προχωρήσει και να προωθήσει αυτό το ζήτημα, ένα ζήτημα το οποίο είναι μεγάλης σημασίας ε, για να προλάβουμε το deadline του 2012. Εμείς σαν πολιτική ομάδα θα συμβάλλουμε σε αυτή την προσπάθεια έτσι που να έχουμε αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό συμφωνώ με εισηγήσεις όπως αυτή που έκανε η κυρία Σίπολ για equal pay for equal work. Είναι το θέμα της πρόσβασης στην αγορά εργασίας και άλλα τέτοια ζητήματα, τα οποία εμείς θα μελετήσουμε με προσοχή και θα επανέλθουμε με συγκεκριμένες τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ. Thank you. Thank you. Now, Mrs. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Χέρστ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για τους φιλελεύθερους, και εγώ μπορώ να πω, ότι το χαιρετίζουμε ότι τώρα έχουμε αυτό το τμήμα των μέτρων από το πακέτο ασύλου που σε βάθος και πιο έντονα θα τεθεί σε διαπραγμάτευση. Σίγουρα είναι κέρια σημασία σημείο να υπάρχει συνεκτικότητα μεταξύ των διαφορετικών οδηγών, να διασφαλίσουμε αυτή τη συνεκτικότητα και συνάφεια. Και στις άλλες οδηγίες αυτό είχαμε πει ότι πρέπει να γίνει. Και για την έννοια της οικογένειας όσον αφορά τον ορισμό, είναι θεμελιώδου σημασία να χρησιμοποιείται ένα ορισμό για το τι εστί οικογένεια, αλλιώ θα υπάρχει πρόβλημα. Τώρα, για την οδηγία, ίσω αυτή είναι μία από τι πιο σημαντικέ και πιο κέρυε, διότι αυτή είναι η οδηγία που επιτόπου θα έχει τη μεγαλύτερη επίπτωση στη ζωή των ανθρώπων. Πού θα στεγάζονται, Ποιο συσίτιο θα παίρνουν, πώς θα τρέφονται, θα παίρνουν κουπόνια, χρήματα, ποια υγειονομική κάλυψη θα έχουν, ποια πρόσβαση στην αγορά εργασία θα έχουν. Όλα αυτά θέματα που πρέπει να προσεχτούν ιδιαίτερα, ώστε όλες αυτές οι πτυχέ της ολοκλήρωσης, της κοινωνικής ένταξη να εντάσσονται ευθύ εξ αρχή στο σωστό πλαίσιο, με σοβαρό τρόπο. Και αν υπάρξει αρνητική έκβαση, δεν θα ήταν του κάκου και δεν θα πάει του ε, στράφη η περίοδος που παρέμειναν αυτοί οι πρόσφυγες ε, τούντες άσυλο ανάμεσά μας. Θα τους έχουμε αντιμετωπίσει με αξιοπρέπεια. Και αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα το οποίο είναι χειροπιαστό και εξειδικευμένο. Και για τους πολίτες, για την κοινή γνώμη είναι ένα πολύ ευαίσθητο, καυτό θέμα. Τα κράτη-μέλη πολύ γοργά και με σαφήνεια είπαν δεν θέλουν πρόσθετες δαπάνες, δεν θέλουν πρόσθετα κόστη. Φοβούνται τα πρόσθετες τις πρόσθετες δαπάνες. Είναι δική μας ευθύνη να εργαστούμε για αυτό το πολύ σοβαρό ευαίσθητο θέμα. Να πούμε τι θα γίνει και τι δεν θα γίνει. Ώστε να μην υπάρξει αναζωπήρωση αρνητικών αισθημάτων από πλευράς μας με τα αποτελέσματα που θα δώσουν. Αν ε, ολοκληρώσαμε τη συζήτηση, να δώσουμε το λόγο στον κύριο Μασίπ. Όπως έλεγα και πριν, εγώ είμαι διαθέσιμος να ακούσουμε δηλαδή και την Προεδρία την... για να μπορέσουμε να λύσουμε τα προβλήματα αυτού του ντοσιέ. Όπως είπε και η βουλευτής του ΕΛΚ, θεωρώ ότι το σύνορο μεταξύ ασύλου και μετανάστευσης είναι ουσιαστικότατη. Όταν θα το έχουμε καθαρό εμείς οι πολιτικοί, τότε μπορούμε να το διαβιβάσουμε και στην κοινωνία για να αποφεύγει τις, συνθήκες, της συγχύσεις. Ένας πρόσφυγας είναι αυτός ο οποίος καταδιώκεται για τις ιδέες του στη χώρα προέλευση και μετά, άμα υπάρχει ελευθερία, πρέπει να δούμε ποιες είναι οι οικονομικές συνθήκες. Αυτό είναι και το προήμιο όλης της ιστορίας, δηλαδή άμα ξεκαθαρίσουμε σαφώς και πούμε ότι εμείς ανεξάρτητα από οτιδήποτε άλλο θέμα που αφορά στην μετανάστευση, εμάς δεν μας ενδιαφέρει η μετανάστευση, μας ενδιαφέρουν οι ετούντε στο άσυλο, αυτοί που διώκονται στη χώρα προέλευσης. και αυτή η όρη είναι εντελώς προσωρινή. Εμένα η οικογένειά μου διώχθηκε στην εποχή του φραγκισμού. Και τότε ο κόσμος έφευγε, αλλά μετά που ήρθε η δημοκρατία δεν άρχισαν να τρέχουν οι Ισπανοί αριστερά-δεξιά ανά τον κόσμο. Εμείς μιλάμε για δύο κόμενους οι οποίοι διώκονται τόσο άγρια που θα λέγαμε ότι υπόκεινται γενοκτονία. Εμείς ως προασπιστές στην Ευρώπη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε αυτό για να τοποθετήσουμε σωστά. Ολοκληρώνουμε τη συζήτηση για αυτό το σημείο. Και πάμε στο επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Δεκαεννέα. Χρησιμοποίηση των προσωπικών ε, στοιχείων των επιβατών. Για το PNR, ο Τίμωθη Κίρκοπ ε, είναι ο εισηγητής μας. Ε, Πρόκειται για μια πρόταση οδηγίας για τη χρησιμοποίηση των προσωπικών στοιχείων επιβατών, ε, για την, ε, τον εντοπισμό ε, και την, τη σύλληψη και την καταδίκη των τρομοκρατών. Δεν θα συζητήσουμε πάρα πολύ το θέμα αυτό, απλώς θα το συζητήσουμε επαρκώς διότι το κείμενο αυτό ε, έρχεται μετά από μια συμφωνία πλαίσιο στο, για τη, στη συνθήκη της Λισαβόνας σε σχέση με τη χρήση του συστήματος PNR των προσωπικών στοιχείων επιβατών τουλάχιστον στις διεθνείς πτήσεις Υπήρξαν πολλές απόψεις που ακούστηκαν από το EDPS, ε, από τον Ευρωπαίο Υπόπτη για την Προστασία Δεδομένων, ε, από την ομάδα εργασίας του άρθρου 29, την ομάδα εργασία του Συμβουλίου, την Υπηρεσία ε, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, όπως επίσης και από την ΕΙΕΔ. Θα μας πει ε, θα μας παρουσιάσει ε, την κατάσταση ο κύριος ε, Κίρκοπ, ενδεχομένω και η Επιτροπή αν το θέλει και μετά θα γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της Επιτροπής. Έχετε το λόγο κύριε Κίρκοπ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πραγματικά πρόκειται για μια ανταλλαγή απόψεων υπαριθμών 1α για να το πω έτσι γιατί έγινε ήδη μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων προσπαθήσαμε εν πάση περιπτώσει να ε, έχουμε μια ανταλλαγή απόψεων, ε, αλλά επειδή ήταν στην ημερήσια διάταξη σε κάποια χρονική στιγμή που έπρεπε να φύγουν πολλοί συνάδελφοι και δεν είχαμε πολύ χρόνο, υποθέτω ότι είναι και η ε, σημερινή κατάσταση η ίδια. Κύριε Πρόεδρε, δεν βλέπω πολλούς συναδέλφους και μπορεί να περάσουμε σε ανταλλαγή απόψεων ένα β ενδεχομένως. Εν πάση περιπτώσει, είναι κάτι για το οποίο δεν περιμένουμε άμεσα αποτελέσματα για να σας πω την αλήθεια. Εγώ σε συγκητής είμαι όσο πιο χαλαρός μπορώ, γιατί πραγματικά ε, πιστεύω ότι δεν θα έπρεπε να βιαστούμε πριν δώσουμε σε όποιον έχει άποψη για το θέμα αυτό, να έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να πει την άποψή του στην Επιτροπή μας, και οι οργανισμοί έχουν απόψεις ε, τις οποίες θα έπρεπε να μας γνωστοποιήσουν. Είναι σημαντικό να ακούσουμε όλες τις απόψεις. Η άποψή μου λοιπόν είναι... Ελπίζω να μην ε, Επειδή εμείς πρέπει, εγώ ως συγητής πρέπει να ε, συντάξω την έκθεσή μου και επειδή αυτή είναι η βάση της ε, συζήτησης στην Επιτροπή και είναι η βάση ε, επί της οποίας πρέπει να ληφθεί απόφαση, ε, και επειδή αυτή τη στιγμή δεν έχω έκθεση στη δια, στη δια, να, σας, προτείνω, ελπίζω να έχω το φθινόπωρο, ελπίζω να είναι επικοδομητική ε, η συνεισφορά ε, των συναδέλφων και να ε, μην προσπαθήσουν να με κάνουν να αποκλίνω από το έργο μου με τις απόψεις τους. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα αυτό ε, είναι ένα ζήτημα που ε, απασχολεί ιδιαίτερα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι δεν είναι παρόντες σήμερα. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία με αυτούς τους συναδέλφους για άλλα ζητήματα που δεν αφορούσαν τα προσωπικά στοιχεία επιβατών, όμως το PNR είναι ένα ζήτημα διαφορετικό ε, σε σχέση με τα άλλα που έχουμε εξετάσει ως σήμερα. Ε, υπάρχουν όμως κάποια στοιχεία τα οποία είναι δύσκολα, πρέπει να τα ελέγξουμε πολύ προσεκτικά και ε, υπάρχουν και ζητήματα που έχουν να κάνουν καθαρά με τα θέματα δεδομένων. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα αυτό. Τα δεδομένα, τα προσωπικά, αθώων ανθρώπων σε, στις περισσότερες περιπτώσεις και γι' αυτό πρέπει να θέσουμε κριτήρια και να δούμε πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα δεδομένα. Πρέπει λοιπόν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποφασίσουμε πόσο, πόσο, θέλουμε, πόσο εκτεταμένη θέλουμε να είναι αυτή η συμφωνία PNR, ποια είναι η έκβαση αυτής της συμφωνίας, ποιος ήταν ο αντίκτυπος, ποιος το χρηματοδοτήσει το κόστος το οποίο προφανώς υπάρχει και ποια θα είναι τα κριτήρια για την τελική χρήση των δεδομένων. Είπα στις παρατηρήσεις μου ότι υπήρξε η εξής κατάσταση όλα όσα λέμε τα βασίζουμε στις προτάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέχρι τώρα. Είχαμε πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις ε, ως τώρα και αναφερθήκατε κι εσείς σε μερικέ από αυτές, από πολλές υπηρεσίες ε, ε τις οποίες γνώριζα από το παρελθόν, ε, υπήρξαν και ορισμένε που δεν τις γνώριζα από εγώ πιο πριν, ακούσαμε τις απόψεις πολλών νομικών και επειδή και εγώ είμαι νομικός θα ήθελα απλώς να ε, κρούσε τον κόδυνα του κινδύνου ε, σε σχέση με τις απόψεις ε, των ομίλων, των, των, νομικών, γιατί ακούσαμε πολλές φορές την άποψή τους και ακούσαμε άλλωστε και από πολλά συνταγματικά δικαστήρια, στη Ρουμανία για παράδειγμα, για την διατήρηση των δεδομένων. Πολύ καλά κάνουν, χαίρομαι πολύ που ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό και θα έχω και εγώ πολλά ερωτήματα προς, εκείν, προς τους προς το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ρουμανία. Θα έχουν και εκείνοι πολλά ερωτήματα προ εμένα σε σχέση με, τις, ε, με τη συλλογή σορευτικών πληροφοριών. Είναι ένα τομέα που θα έπρεπε όντω να μας απασχολήσει και θα ήθελα να ασχοληθώ ειδικότερα με αυτό το θέμα. Θα ακούσουμε βέβαια και άλλες απόψεις, όπως για παράδειγμα ε, από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Του ζήτησα να περιμένουν για τις παρατηρήσεις τους, για ε, την έκθεσή μου και δέχθηκαν την ε, πρόταση αυτή. Πιστεύω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούσω τις παρατηρήσεις ε, για την έκθεσή μου. Θα είναι πιο ενδιαφέρουσες από τις παρατηρήσεις που έχω λάβει ως τώρα για την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι για την δική μου έκθεση. Κάτι ακόμη θα ήθελα να πω. Έχει μόλις αρχίσει η δουλειά επί του θέματος αυτού. Εγώ πιστεύω πραγματικά ότι υπάρχει ανάγκη ύπαρξη συμφωνίας. Δεν θα αρχίσει τη δουλειά αυτή ο συζητητή αν δεν πίστευα κάτι τέτοιο και κατά την άποψή μου το PNR είναι ένα πάρα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την καταπολέμηση ε, των σοβαρών ε, οργανωμένων εγκλημάτων και της τρομοκρατίας. Ξέρω ότι αναμοχλεύει διάφορα ε, αισθήματα μεταξύ των μελών της Επιτροπής μας και έχουν το δικαίωμα να πούν ό,τι θέλουν βεβαίως, αλλά νομίζω ότι είναι, πρέπει, πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβουμε την ευθύνη, να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε ε, αυτούς τους αθώους ε, ταξιδιώτες αλλά και τους αθώους πολίτες όσο καλύτερα μπορούμε. Ε, εξισορροπώντας βέβαια την ανάγκη της ιδιωτικότητάς τους και της προστασίας των δεδομένων. Όλα αυτά τα έχω στο μυαλό μου κύριε Πρόεδρε όταν αρχίζω το ταξίδι της έκθεσης αυτής και ε, ελπίζω ότι μπορώ να βασιστώ και στην συνεργασία των συναδέλφων και στη δική σας συνεργασία κύριε Πρόεδρε και ελπίζω να καταλήξουμε σε ένα πολύ ικανοποιητικό αποτέλεσμα. Και την επόμενη φορά που θα συζητήσουμε το θέμα αυτό θα είναι το φθινόπωρο και ε, αναμένω εναγωνίω την ευκαιρία αυτή. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κύρκοφ. Έχετε δίκιο, δεν είναι η πρώτη φορά που είχαμε μία πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Μετά έχουμε μία ε, ανταλλαγή απόψεων ένα α, ένα β, ένα γ και ούτω καθεξής. Και όπως είπατε ε, κύριε Κύρκοφ, ε, Ελπίζω ότι η παρουσίασή σας ε, είναι μια καλή βάση για ε, επικοδομητική για επικοδομητικές παρατηρήσεις ε, ε, από τους συναδέλφους. Ελπίζω αυτή να είναι η περίπτωση και όχι αντίθετη. Ε, δεν ξέρω αν εκπρόσωπο Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλει να πάρει το λόγο, ο κύριος Ζούνιος Αλμέιδα και μετά το Συμβούλιο. Πριν αρχίσει η συζήτηση με τα μέλη της Επιτροπής. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Θα εξοικονομήσω το χρόνο σας, Πρόεδρε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη παρουσιάσει τις προτάσεις της. Δεν θα ήταν χρήσιμο, πιστεύω, να τις ξαναπαρουσιάσω εγώ. Βρισκόμαστε εδώ να ακούσουμε τις δικές σας απόψεις, τι έχετε εσείς να μας πείτε. Και θα είμαστε έτοιμοι να δώσουμε απαντήσεις στις ερωτήσεις μας σχετικά με αυτά. Σε αυτή τη φάση όμως δεν έχω τίποτα να προσθέσω. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε κύριε. Για την Πολωνική Προεδρία θα λάβετε τον λόγο παρακαλώ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχηθώ ένα πολύ καλό απόγευμα σε όλους τους Ευρωβουλευτές στο Σώμα, στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Θα ήθελα να ήμουν και εγώ σε θέση, όπως και ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να πω ότι το κάναμε στο παρελθόν, αυτό το καλύψαμε. Κατά κάποιο τρόπο το καλύψαμε στο παρελθόν. Προτού έρθω τώρα στις λεπτομέρειες της θέσης της Πολωνικής Προεδρίας για αυτό το θέμα σήμερα σε σχέση με το PNR, με τα θέματα των προσωπικών δεδομένων ταξιδιωτών, να σας δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία. Πρώτον, είναι η τρίτη διατύπωση αυτής της πρότασης, αυτή που έχουμε μπροστά μας. Και υποθέτω ότι θα έπρεπε να κάνουμε ό,τι γίνεται καλύτερο, ώστε να μην ακολουθήσει η τέσσερα αν θυμάμαι καλά, είναι η πέμπτη ή έκτη προεδρία από τον καιρό όχι ξαναξεκινώντας, αλλά συνεχίζοντας τη δουλειά στο ίδιο αυτό χαρτοφυλάκιο. Και δεν είναι όλο και πιο εύκολα τα πράγματα, αλλά το αντίθετο περιπλέκονται. Σε αυτή τη χρονική στιγμή και σε αυτή τη συγκυρία θέλω να ευχαριστήσω τους ε, προηγούμενους και τους ε, ε, για την κατεύθυνση που δόθηκε σε σχέση με αυτά τα θέματα και που θα συνεχίσει η Πολωνική Προεδρία προς αυτή την κατεύθυνση. Τρία σημεία θέλω να αναφέρω. Το πρώτο, το περιβάλλον στο οποίο ξεκινήσαμε το έργο μας. Το δεύτερο, ο στόχος που ταπεινά επιθυμούμε και ελπίζουμε θα επιτύχουμε. Το τρίτο, η λύση. Η λύση που αυτή τη στιγμή μπορώ μόνο γενικόλογα να αναφέρω, αλλά κατανοώ ότι αν είμαστε αφελείς και υπερ, ε, υπερ φιλόδοξοι, δεν θα καταφέρουμε να πετύχουμε έναν πραγματικό συμβιβασμό που να είναι αποτελεσματικός μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Για τη λύση, να πω ότι υπό τη συναπόφαση ε, θα ληφθεί. Δεν μπορώ κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας μου να βρω ένα πιο χαρακτηριστικό και δύσκολο παράδειγμα νομοθεσίας για το δυσχερές του χαρακτήρα της συμφωνίας, για το περιβάλλον. Θα ήθελα να πω ότι ακριβώς αυτή η δυσκολία αυτού του φυλακίου απαιτεί και αξίζει υπομονή, αποσαφήνιση των θεμάτων και προσπάθεια να βρούμε εξειδικευμένε, στοχοθετημένε προτάσει. Και θα ήθελα να συμμεριστώ μαζί σα τι απόψει για το χρονοδιάγραμμα. Είχαμε την πρώτη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των κρατών μελών και ε, τη ομάδα εργασία για την γενική αξιολόγηση. Στι θερινέ διακοπέ στοχεύουμε να βρούμε να έχουμε συγκεκριμένε παρατηρήσει που θα θέλαμε το Σεπτέμβριο να ληφθούν υπόψη. Τέλη Σεπτεμβρίου θα επανέλθουμε προ τα κράτη-μέλη για επανεξέταση. Μια κέρια σημασία πληροφορία που θα ήθελα να σημειώσετε κυρίε και κύριοι. Ποτέ δεν θα καθυστερήσουμε στο να έρθουμε σε επαφή μαζί σα. Όχι για θέματα πολιτική ορθότητα, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι αν δεν μπορεί να επιτευχθεί μια τελική λύση, αν δεν συζητούμε ο ένα με τον άλλο για το στόχο μα, δεν θα το πετύχουμε. Στο πρώτο έγγραφο που παρουσίασε στην ομάδα εργασίας η Πολωνική Προεδρία, ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη και μπορώ να είμαι πιο ε, πλήρης και ενημερωτικός πρέπει να βρεθούν απαντήσεις στα ερωτήματα με την αναλογικότητα και την αποτελεσματικότητα και με τον κίνδυνο να επαναλάβω τον εαυτό μου ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να υποβάλουν τις προτάσεις τους προς την Πολωνική Προεδρία. Να βρούμε μια κοινή γλώσσα για τη διατύπωση που θα μπορέσει να ενταχθεί στο κείμενο. Δεν θέλω να υπάρξει ανάμειξη με το προήμιο όπως πολύ συχνά γίνεται. Προσπαθούμε να βρούμε μια λύση που ουσιαστικά θα κλείσει για τα κράτη-μέλη που βρίσκονται πιο απομακρυσμένα από τη συνένεση αυτά τα θέματα σε σχέση με το διάλογο, τη διαβούλευση τελευταίο σημείο, λύση. Αν εργαστούμε και συνεργαστούμε από κοινού με διαφάνεια για επίλυση, λάβουμε υπόψη τις παρατηρήσεις των άλλων, μπορούμε να καταλήξουμε σε ένα συμβιβασμό, σε μια λύση. Όχι μόνο με την ομάδα εργασίας, αλλά και με την Επιτροπή ΚΑΤΣ και να επανέλθουμε στο Ευρωκοινοβούλιο να ενημερώσουμε πώς έχουν τα πράγματα. Η τελευταία μου παρατήρηση υποτίθεται ότι θα είναι απόδειξη για την κατεύθυνση που υιοθετήσαμε ως προσανατολισμό. Συνήλθαμε, συναντηθήκαμε κατά την πρώτη συνάντηση της ομάδας εργασίας στις 7 Ιουλίου. Αφιερώσαμε τον περισσότερο χρόνο μας ακούγοντας, αφουγκραζόμενοι, όχι ο, παρεμβαίνοντας, ομιλώντας εμείς οι ίδιοι. Και έτσι λοιπόν σε σχέση με τα θέματα PNR των ταξιδιωτών να αν συμμεριστούμε απόψει τι είχε γίνει και ποια ήταν η έκβαση. Οι εκπρόσωποι του Ηνωμένου Βασιλείου, της Σουηδίας, της Γαλλίας και του Βελγίου ήρθαν και συμμετείχαν σε, αυτές, σε αυτήν την ανταλλαγή απόψεων. Στη συνέχεια άλλαξε το περιβάλλον. Η ΑΙΑΤΑ, ε, Διεθνή Ένωση Αέριων Μεταφορών, η ε, ο Ευρωπαϊκός Σύλλογος και Ένωση ε, Ταξιδιωτικών Πρακτόρων και οι ταξιδιωτικέ εταιρείε, οι εκπρόσωποι των εταιρεών μίλησαν και έκαναν παρατηρήσει. Οι παρατηρήσει αυτέ θα ληφθούν υπόψη από την Πολωνική Προεδρία σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τέλο, αλλά εξίσου σημαντικό, δόθηκε ο λόγο στην ομάδα εργασία του άρθρου 29 και υπήρξε υπόσχεση δέσμευση τη ΕΚΟΣΟΚ, του εισηγητή από την ΕΚΟΣΟΚ, να επανέλθει το Σεπτέμβριο και να εκφράσει τι απόψει αυτού του ε, πολύ σοβαρού μέλου. Αλλά σε σχέση με τι ενέργειε μεταφορέ, ε, όταν έχουμε τα ψηφί, τις ψηφίδες ε, στο τραπέζι και δημιουργήσουμε την τελική εικόνα στο παζλ, πρέπει να είμαστε σε θέση να προτού ολοκληρωθεί η δουλειά, πρέπει να δούμε και να αποδείξουμε ότι ζητήθηκε από τον κάθε ένα να εκφράσει τις να εκφράσει τις απόψεις του και να είμαστε ε, πλήρεις ε, στη δουλειά μας, ώστε να είναι γνωστό πού βρίσκεται το Συμβούλιο, να γνωρίζουμε ποια θέματα κάλυψαν και με ποιο τρόπο παρενέβησαν, να μην υπάρξει κάποια παρανόηση, να είναι μια καλή πρόταση που πρέπει να τελειοποιηθεί και να εγκριθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ήσασταν πάρα πολύ ειλικρινείς. Νομίζω ότι έχουμε... Έχει αυτή τη στιγμή να ανοίξουμε την ε, συζήτηση τώρα. Η κυρία Σίπερ πρώτη. Λυπούμε που τόσο συχνά παρεμβαίνω σήμερα. Δεν υπάρχουν πολλά μέλη, γι' αυτό ζήτησα να παρέμβω πάλι. Έχετε το δικαίωμα, είναι απόλυτο δικαίωμά σα, κυρία, λέει ο πρόεδρο. Θα ήθελα με ένα θέμα θεμελιώδου σημασία, αρχή, ένα θέμα αρχή να ξεκινήσω. Ξέρω ότι δεν το εννοούσε έτσι η Προεδρία του Συμβουλίου, αλλά ω θέμα αρχή θέλω να πω μια οδηγία μόνο έτσι να εγκριθεί, επειδή υπήρξαν αρκετέ προσπάθειε στο παρελθόν και απέτυχαν, είναι κακό επιχείρημα. Δεν είναι πιστικό. Πρέπει να δούμε δούμε ποια είναι η πρόσθετη αξία, το πρόσθετο αποτέλεσμα που προσφέρει η οδηγία. Αν επανειλημμένα απέτυχε στο παρελθόν, ε, τότε να σκεφτούμε τι χρειαζόμαστε καν. Αλλά ακόμα και οι όροι προσέγγισης και οι όροι πλαίσιο, πλαισίου υπό τους οποίους συζητείτε, πραγματικά δηλαδή χρειάζεται χρόνος για τη συζήτηση, γι' αυτό η προσέγγιση του Timothy Kirkhope είναι σωστή. Προσεκτικά όλα τα σημεία να τα αναλύσουμε και να τα συζητήσουμε. Πολύ λογικό αυτό. Αν καταλήξουμε στο συμπέρασμα αυτή η οδηγία δίνει πρόσθετη αξία και αποτέλεσμα για την καταπολέμηση του σοβαρού οργανωμένου εγκλήματος, ε, τότε αμέσως τίθεται το ερώτημα στη συνέχεια της υλοποίησης ε, της ε, εκτέλεσης, της αρμοδιότητας. Ποιος θα έχει πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, σε αυτή την κοινότητα των 27 κρατών μελών. Ένα κράτος μέλος θα είναι αρμόδιο για συγκεκριμένο έργο, από κοινού θα τα διοργανώσουμε. Ποιος θα έχει πρόσβαση, ποιος θα συλλέγει αυτά τα στοιχεία, τα προσωπικά δεδομένα. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πολύ, πολύ μεγάλη σημασία, όπου έχουμε και αντιπαράθεση και σε σχέση και με τη Διεθνή Συμφωνία για τα δεδομένα των ταξιδιωτών, όπου απαιτείται να, για να καταλήξουμε σε μια συμφωνία να πετύχουμε την υλοποίηση των δικών μας αιτημάτων έναντι τρίτων, έναντι συμβαλωμένων μερών. Τα αιτήματά μας να είναι σεβαστά, στις διεκδικήσεις μας και για τους στόχους και για τον ορισμό όχι μόνο τρομοκρατίας αλλά και τον, οργανισμό, τον ορισμό οργανωμένου εγκλήματος πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί να μην υπάρχει κίνδυνος κάποτε όλα αυτά τα στοιχεία να χρησιμοποιούνται και για τα πιο μικρά δικήματα ή παραπτώματα και έτσι να είμαστε υπερβολικοί. Δεν θα μπορούμε με τέτοιο τρόπο να υπερβάλλουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ίνιτφελτ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς ε, να ζητήσω συγγνώμη γιατί θα πρέπει να φύγω μετά από την παρέμβασή μου. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την, ε, το πολύ ανοιχτό πνεύμα και τη μέθοδο εργασίας ε, που ακολουθεί. Νομίζω ότι είναι ένα σίγουρος τρόπος για ένα καλό αποτέλεσμα και μια καλή συνένεση. Πρέπει να είμαστε πολύ ρεαλιστές όμως νομίζω για το θέμα αυτό πρέπει να δώσουμε στις μηχανισμούς επιβολής του νόμου τα μέσα για να διεκπαιρεώσουν τα καθήκοντά τους. Τίποτε παραπάνω, τίποτε λιγότερο. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς στην τοποθέτησή μας. Ό,τι αποφασίσουμε πρέπει να βασίζεται σε στοιχεία και αυτό είναι κάτι το οποίο μέχρι τώρα δεν έγινε. Ξέρω ότι η Πολωνική Προεδρία συμφωνεί απολύτω με αυτό, αλλά περιμένουμε ακόμη, παρά το γεγονός ότι έχουμε κάποιες πληροφορίες τουλάχιστον από τον εισηγητή και από την παρουσίαση που οργάνωσε ο ίδιος στο Μάντσεστερ, το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να ε, δούμε κατά πόσο υπάρχει ε, τόσο μεγάλη ανάγκη, τόσο ε, ευρεία συλλογής πληροφοριών. Αυτό πρέπει να δούμε κατά πόσο χρειάζεται ή όχι και είναι πραγματικά δύσκολο να δείξουμε κατά πόσο είναι αναγκαίο αυτό. Πρέπει όμως για να το κάνουμε να κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που κάναμε ως τώρα. Πρέπει επίσης να καταδείξουμε την αναγκαιότητα για ένα πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Ένωσης για το PNR, γιατί η άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν κάποτε, αν δεν το κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα έχουμε ένα, ε, μια επικόλυση των 27 διαφορετικών συστημάτων και ε, υπάρχει ένα μόνο το οποίο λειτουργεί πλήρως και αυτό είναι το Βρετανικό. Υπάρχουν κράτη-μέλη που λένε ότι κάτι κάνουν, όπως και το δικό μου κράτος μέλος, επισήμως όμως δεν συλλέγουν PNR, όμως το κάνουν επί τη βάση ε, μίας ε, καθόλου στέρεας νομικής βάσης. Οπότε ε, το λέω αυτό επί τη ευκαιρία. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει νομικά μία υποχρέωση να γίνεται κάτι τέτοιο. Ε, χρειαζόμαστε ένα πολύ σαφώς ορισμένο πεδίο εφ, εφαρμογής και κάτι ακόμη, και με αυτό θα ολοκληρώσω, πιστεύω ότι είναι όμως πολύ σημαντικό είναι το ζήτημα της ε, μακροχρόνιας αποθήκευσης των δεδομένων, όλων των δεδομένων. Γιατί αυτό που κάνουμε δεν είναι ότι χρησιμοποιούμε απλώς τα δεδομένα για να παρακολουθήσουμε όσους περνούν ε, κάποιο σύνορο, γιατί αυτό είναι το λιγότερο προβληματικό στοιχείο. Το πιο προβληματικό στοιχείο είναι ότι αποθηκεύουμε μαζικά δεδομένα αθώων ανθρώπων για εγκλήματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, εν πάση περιπτώσει για δικήματα που δεν έχουν γίνει καν ακόμα, που δεν έχουν διαπραχθεί και Γι' αυτό ίσως θα πρέπει, ε, δίνουμε και τη δυνατότητα μάλιστα σε μερικού έχουν πρόσβαση σε αυτά τα δεδομένα χωρί δικαστική εντολή. Αν κάποιο δηλαδή θέλει να έρθει και να ερευνήσει το σπίτι μου, θέλει ένταλμα. Δεν μπορεί να μπει μέσα στο σπίτι μου και να αρχίσει να ψάχνει. Οπότε, γιατί επιτρέπουμε να κάνει κάτι τέτοιο κάποιο σε μια βάση δεδομένων προσωπικών στοιχείων κάποιων ανθρώπων. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό δεν μιλούμε μόνο για μια τεράστια βάση δεδομένων αρχείων επιβατών, ε, γιατί δημιουργούμε και μία βάση δεδομένων, τραπεζικών δεδομένων, τηλεπικοινωνιακών δεδομένων και στο τέλος θα έχουμε τεράστιες βάσεις δεδομένων ε, ε, εκατομμυρίων πολιτών που δεν έχουν κάνει τίποτα και ποτέ μπορεί, μπορεί και να μην κάνουν και ποτέ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Άλμπρεχτ. Ο κύριος Άλμπρεχτ, ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. <coughs> το βρίσκω σωστό και σημαντικό τόσο πρόημα, τόσο έγκαιρα να εξετάζουμε αυτή την πρόταση και ευχαριστώ τον κύριο Κέρκοπ για το ότι έχει, έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν και συνεχίζουμε να συζητάμε με βάση το έργο που έχει επιτελέσει. Αυτό είναι σημαντικό και η προσέγγιση είναι και σωστή και αυτή νομίζω. Είναι απόλυτα σημαντικό και όλοι συμφωνούμε σε αυτό η τρομοκρατία και το έγκλημα, το οργανωμένο έγκλημα να καταπολεμηθούν. Και είναι απόλυτα αναγκαίο οι αστυνομικέ αρχέ και οι δικαστικέ αρχέ να εξοπλιστούν με τα αναγκαία μέσα και εργαλεία για τι ανακρίσει, διακριβώσει, έρευνε για του υπόπτου και να συλλέξουν στοιχεία. Αυτό για το οποίο κάνουμε λόγο εδώ είναι ένα μέτρο το οποίο πιο πριν ξεκίνησε και ξεκινά και ξεκινά όταν δεν υπάρχει ακόμα υποψία ή συγκεκριμένη έρευνα εις βάρος κάποιου. Σημαντικό είναι να το πούμε αυτό και έχουμε κάποιες επικρίσεις που διατυπώθηκαν και ακούστηκαν. Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις επικρίσεις και τις γνωμοδοτήσεις που άκουσα και τις απόψεις που άκουσα πρέπει να πούμε με σαφήνεια ότι η πρόταση που έχει υποβληθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είναι αναλογική, δεν είναι αποδεκτή δεν είναι αυτό αποδεκτό. Πρέπει να το πούμε ξεκάθαρα. Σταράτα, ε, κοφτά, ορθά κοφτά. Δεν είναι ουσιαστικά η σωστή βάση αυτή. Αποθήκευση πέντε ετών διάρκειας όλων των προσωπικών δεδομένων Ευρωπαίων πολιτών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο. Αυτό είναι κάτι δυσανάλογο, πραγματικά υπερβολικό και δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Απλά και μόνο επειδή η σημερινή χρήση των στοιχείων των ταξιδιωτών από διαφορετικά κράτη σήμερα έχει τελείως διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις. Για τελείως διαφορετικούς στόχους χρησιμοποιούνται, διαφορετική διάρκειας και δεν υπάρχει συμφωνία αν αυτά τα στοιχεία αποκλειστικά για την καταπολέμηση τρομοκρατίες θα χρησιμοποιούνται ή αποκλειστικά για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Το ότι δεν συμβαίνει αυτό σε ενιαίο πλαίσιο το βλέπουμε στις συμφωνίες που διαπραγματευόμαστε με τρίτες χώρες. Υπάρχουν πολύ σημαντικά ερωτήματα. Η μακροχρόνια αποθήκευση έχει αναφερθεί. Γιατί είναι αναγκαία αυτή. Γιατί για παράδειγμα <coughs> η ανάλυση του οργανωμένου έγκληματος δεν μπορεί με ανώνυμο τρόπο να οδηγήσει στη συλλογή δεδομένων ανώνυμα χωρίς ε, ε, γιατί δεν μπορούν κλασικές μέθοδοι έρευνας ε, να ενισχυθούν όπου η συγκεκριμένη δουλειά των αστυνομικών αρχών στα αεροδρόμια και εκεί όπου υπάρχουν γεγονότα συμβάντα όσον αφορά το οργανωμένο έγκλημα διότι αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Κάνουν οικονομίες, εξοικονομούν σε σχέση με το έργο της αστυνομίας, σε σχέση με τις ανακρίσεις και ε, έρευνες και στο τέλος τέλος υποβάλλουν τέτοιες προτάσεις που είμαστε πεισμένοι ότι δεν θα είναι αποτελεσματικές. Στο τέλος τίθεται το, το θέμα της συνταγματικής συμβατότητας και της συμβατότητας με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μιας τέτοια πρότασης. Πρέπει να το δούμε υποχρεωτικά. Μια τέτοια δυνατότητα είναι συμβατή με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι δυνατό να γίνει κάτι τέτοιο. Και τα όσα νομικά είδαμε για την ποιότητα των νομικών γνωμοδοτήσεων μπορεί κανείς να έχει διαφορετικές απόψεις. Όπου υπάρχουν δύο νομομαθείς υπάρχουν δύο διαφορετικές απόψεις. Σαφές αυτό. Αλλά οι σαφές επικρίσεις, ε, σαφείς επικρίσεις έχουν ήδη διατυπωθεί από ειδικού δίκαστες, νομομαθείς. Δεδομένης μιας τόσο διαφορετικής κατάστασης δεν είναι δυνατόν να μην λέμε ούτε λέξη όπως κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για όλα αυτά τα πράγματα. Αυτό είναι πραγματικά δυσνόητο, είναι απαράδεκτο. Έχουμε ένα συνταγματικό πλαίσιο. Υπάρχει ερώτημα. Πού σταματάει η διαχωριστική γραμμή αυτή την αποθήκευση και διαφύλαξη στοιχείων προσωπικών δεδομένων των πολιτών. Δεν θα είναι δυνατόν οι πολίτε μα να τα δεχθούν όλα αυτά αν δεν τραβήξουμε σαφεί διαχωριστικέ γραμμέ που είναι τα όρια όλων αυτών των δράσεων. Ευχαριστώ. Mrs. Ernst. Κυρία Ernst, παρακαλώ. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ. Ξεκινώντας έτσι, πρέπει να πω ευθύ εξ αρχή είχαμε μεγάλες αμφιβολίες. Μεγάλες αμφιβολίες ότι τέτοιου είδους συμφωνίες όπως για το PNR, για τα προσωπικά δεδομένα ταξιδιωτών έχουν νόημα. Πουθενά δεν υπάρχει απόδειξη ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και πρέπει να γίνεται και από την άλλη πλευρά και τα επιχειρήματα που η ίδια η Επιτροπή χρησιμοποιεί και που η ίδια στην πρότασή της αναφέρει δεν είναι πιστικά, δεν ευσταθούν. Και το επιχείρημα ότι κάποια κράτη θέλουν, επιθυμούν να έχουν τέτοιες ρυθμίσεις δεν αποσαφηνίζονται με τέτοια επιχειρήματα τα πράγματα και δημιουργούνται σημαντικές δυσκολίες έτσι. Και δεν είναι μόνο οι επικρίσει οι δικέ μα, αλλά και η ίδια η Υπηρεσία για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα έχει μια εξοντοτική κριτική που διατύπωσε ει βάρο τη μη αναλογικότητα αυτού του μέτρου, αυτή τη πρόταση. Και ρωτά και εκείνη ποιο είναι το νόημα και ποια είναι η χρησιμότητα όλων αυτών όταν παραβιάζονται τα θέματα της αναλογικότητας με τέτοιο έκδηλο ε, ε, τρόπο και πρέπει ειλικρινά να ομολογήσουμε και να πούμε ότι πρέπει να συζητήσουμε ανοιχτά, για παράδειγμα, για τον κατάλογο των αδικημάτων και παραπτωμάτων. Αναφέρεται εδώ καταπολέμηση τρομοκρατίας. Δεν αναφέρομαι σε αυτό. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψη ε, στο εδάφιο 2. Τεράστια απαρίθμηση όλων των άλλων στοιχείων. Εμπρισμό, ε, απάτη, εκβιασμό. πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε λόγο Αυτά εννοούμε ουσιαστικά. Αυτό είναι το νόημα. Αν μια τέτοια ρύθμιση θέλουμε να υπάρξει για τα PNR, για τα προσωπικά δεδομένα ταξιδιωτών και να φτάσουμε τόσο μακριά, είναι πραγματικά προβληματικό. Και μετά έχουμε και την απαγόρευση επεξεργασία συγκεκριμένων στοιχείων όσον αφορά κάποια άτομα. Εδώ στο άρθρο 4 στην πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής σε αυτό αναφέρεται. Γιατί η αρνητική διακριτική μεταχείριση ή η επιλεκτική μεταχείριση. Εδώ λείπει το θέμα του του, της ηλικία, του φίλου, Απόλυτα ελλειπής, ας το πω έτσι, απαρίθμηση ή ε, κατάλογος. Τι θα κάνουμε ή θα συνεχίσουμε με ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Τι γίνεται με τα στοιχεία που αφήνουν να υποθέσει κανείς ότι υπάρχει μια έμεση ή μια διακριτική, έμεση διακριτική μεταχείριση ή επιλεκτική διακριτική αρνητική μεταχείριση. Γιατί όλα αυτά πρέπει να γίνουν. Γιατί αυτά τα, αυτή, μια κεντρική υπηρεσία θα συλλέγει όλα αυτά τα στοιχεία και θα τα αποθηκεύει δεν είναι δεδομένη η αρνητική διακριτική μεταχείριση. Τουλάχιστον αυτό υποψιαζόμαστε και υποθέτουμε. Πώς μπορεί να αποκλειστεί αυτή. Πραγματικό ένιγμα αυτό. Γρίφος. Και σε σχέση με τα κράτη-μέλη. Πραγματικά περίεργη η διατύπωση που επελέγει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν ακολουθηθεί έτσι όπως την προτείνουν. Δεν μπορούμε εμείς να τη δεχτούμε έτσι. Πολλά αναφέρθηκαν για την πενταετή αποθήκευση πενταετούς διάρκειας. Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει γιατί και πώς πρέπει να γίνει αυτό. Πολύ δύσκολο να κατανοήσουμε. Και τελευταίο ένα σημείο θέλω να επισημάνω ακόμα. Για το άρθρο 11 όπως έχει εδώ προστασία προσωπικών δεδομένων και σε σχέση με την νομική βάση για την απόφαση του 2008 ως πλαίσιο ουσιαστικά θα πρέπει να προσανατολιστούμε να δούμε τι θα γίνει στο τέλος τέλος αν έχουμε μια τέτοια ε, βάση και μια τέτοια πρόταση. Αυτό που θα έχουμε θα είναι μια νέα οδηγία για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Μα θέλουμε όμω να εργαστούμε πρώτα για αυτή τη νέα οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα και όχι να την έχουμε κομμένη και αεραμένη μπροστά μα. Α αναμείνουμε λοιπόν να την έχουμε πρώτα αυτή και να μην κάνουμε μισά τα πράγματα ατελή και αν, χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και να, χωρίς να είναι ικανοποιητικά. Βήμα προς βήμα θα πρέπει τα επιμέρους σημεία να τα συζητήσουμε. Αυτό θα ήθελα να γίνει από του σκιώδεις εισηγητές και με τον εισηγητή να έχουμε επαρκή χρόνο ώστε να ξεκινήσουμε και να κάνουμε δουλειά η οποία θα είναι παραγωγική και όχι αντιπαραγωγική μέσα σε αυτούς τους όρους. Ευχαριστώ. Λατφόρντ, your turn. Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ κυρία Λάτφορντ. Um, yes, I... I, I have considerable worries about... Κοιτάξτε, εγώ έχω σοβαρές ανησυχίες για αυτή την πρόταση. Ο όγκος των δεδομένων με απασχολεί και ειδικότερα το γεγονός ότι αφορά κυρίως ε, ε, για τον όρο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άγνωστη ύποπτη. Μα ένας άνθρωπος δεν είναι ύποπτος αν δεν υπάρχει σοβαρή βάση για να είναι ύποπτος. Δεν ξέρει κανείς ε, από την αρχή αν είναι ύποπτος ή όχι. οπότε εγώ δεν συμφωνώ πάρα πολύ με την ιδέα αυτή. Όπως δεν μου αρέσει και ο όρος προφίλ για τα ευαίσθητα δεδομένα προφίλ ταξιδιώτη. Τι θα πει αυτό. Δεν ξέρω. Είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να είχε διαπράξει ένα δίκημα. Δεν λέω ότι δεν, θα είναι, ότι δεν είναι χρήσιμο. Ε, απλώς... Ε, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι χρήσιμο στην, στο εμπόριο ναρκωτικών, ε, στην ε, σωματεμπορία. καταλαβαίνω ότι θα είναι χρήσιμο σε τέτοιου είδους τομείς, αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που πρέπει όλα αυτά τα δεδομένα να διατηρούνται και να αποθηκεύονται ε, για ανθρώπους που είναι αθώοι ή τέλο πάντων που τεκμέρονται αθώοι μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ύποπτοι, πολλό δε μάλλον ένοχοι. Αυτό λοιπόν μου δημιουργεί εμένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι ότι γίνεται όλη αυτή λοιπόν η συλλογή των δεδομένων, υπάρχουν και όλε αυτέ οι προτάσει γύρω από αυτό το θέμα, και εγώ μπορώ να μιλήσω μόνο για τη δική μου χώρα. Αυτή η κουλτούρα της παρατήρηση, της, ε, του σεβασμού των ε, υψηλών επιπέδων ιδιωτικότητας και προστασίας των δεδομένων ε, τελικά δεν υφίσταται. Θα υπάρχει ένα, και μάλιστα ξέρετε ότι υπάρχει και ένα τεράστιο σκάνδαλο στο Ηνωμένο Βασίλειο, πάρα πολύ πρόσφατο, σε σχέση με υποκλοπές, στο οποίο ε, συμμετείχαν δημοσιογράφοι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, ε, ε, υπάρχουν τεράστιες ποινές για αδικήματα που αφορούν την προστασία των δεδομένων ειδικότερα. Και γι' αυτό ακριβώς ανησυχώ. Η αστυνομία παρέχει από τις βάσεις δεδομένων της ε, ε επιχρήμαση ε, ε, προσωπικά δεδομένα ανθρώπων. Και αυτό μας λέει ακριβώς ποια είναι η κατάσταση αυτής της κουλτούρας για την προστασία των δεδομένων και για την πρόσβαση στα δεδομένα. Οπότε, πρόκειται δεν, δεν ξέρω κατά πόσο είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Εντάξει, μπορώ να πιστώ ενδεχομένως ότι είναι χρήσιμο αυτό που συζητούμε κυρίως για τη σωματεμπορία, για το εμπόριο ναρκωτικών, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αναλογικό. Και αυτό ακριβώς ε, είναι αυτό ε, το οποίο θα προσπαθήσει να μας εξηγήσει ο κύριος Κύρκοπ, γιατί πραγματικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δεν έχω δει νομίζω συγκεκριμένα στοιχεία που να δείχνουν ότι το PNR συνεισέφερε στην παρεμπόδιση ή στη σύλληψη ε, ε, τρομοκρατών ενδεχομένω μπορεί να μην έχω ψάξει στο σωστό σημείο για να βρω τα στοιχεία αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχουν τέτοιου είδου παραδείγματα. Δεν γνωρίζω να έχει καταδειχθεί εν πάση περιπτώσει η αναγκαιότητα ύπαρξη των προσωπικών αυτών στοιχείων επιβατών. Ε, μπορώ βέβαια να δω κατά πόσο υπάρχουν πρακτικές εγγύησεις όσον αφορά την ασφάλεια των δεδομένων, το ξέρω ότι το γράφει και η οδηγία αυτό με πολύ γενικό τρόπο ε, ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας για τα προστασία των δεδομένων ε, και σοβαρές ποινές σε περίπτωση παραβίαση των αρχών αυτών. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να φτάσουμε μέχρι το να κλειδώνονται ορισμένα δεδομένα ή, εν πάση περιπτώσει, να υπάρξουν κάποιες όντω πρακτικές εγγυήσεις ότι δεν θα γίνει κάτι τέτοιο. Και για να ολοκληρώσω, με ένα κομπλιμέντο προς τη χώρα μου που τουλάχιστον ε, έχει νομοθεσία για την ε, συλλογή ε, δεδομένων. Εντάξει, χρησιμοποιεί βέβαια τη λέξη profiling, αλλά ενδεχομένως να είναι πιο κρίσιμος αυτός ο όρος ε, από το να καθόμαστε να συζητούμε, ε, να ψάχνουμε όρο για να το πούμε και η κυρία Ίνετφελντ άλλωστε μίλησε για το γεγονός ότι δεν υπάρχει στέρεα νομική βάση στη δική τη χώρα τουλάχιστον το Ηνωμένο Βασίλειο το κάνει με έναν τρόπο απολύτω εμφα... απολύτως εμφανή και σαφή αυτό. Κύριος Τριανταφυλλίδης. Πρόεδρε, συμμερίζομαι τι περισσότερε απόψει που εκφράστηκαν από την κυρία Λάντφορντ και από την προλήσασα. Όμω δεν θα σχολιάσω τι προτάσει τη Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί όπω είπε ο εισηγητή, είναι η δική του έκθεση. Από πλευρά τη πρέπει να υπάρξουν σχόλια και αξιολογήσει, και έτσι πρέπει να προχωρήσουμε. Σε αυτή τη φάση θέλω να πω ότι όπως και σε άλλες περιπτώσεις που αφορούν την επιβολή των νόμων και εδώ στα προσωπικά δεδομένα ταξιδιωτών είναι η εξέβρεση της σωστής ισορροπίας μεταξύ της ανάγκης να επιβληθεί ο νόμος και της διαφύλαξης και προστασίας των προσωπικών δικαιωμάτων. Προσβλέπω στην προσέγγιση του εισηγητή και θα αναμείνω ώστε να υπάρξει έκθεσή του και με αποκοινούμε τον εισηγητή και τους άλλους σκιώδεις να συζητήσουμε για την επίτευξη των ευκταίων αποτελεσμάτων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τώρα, πρωτού επανέλθω σε κύριε ε, Κέρκοπ. Ο κύριος ε, Νούνες Αλμέιδα τώρα θα ήθελε να αναφέρει κάτι. Αν επιθυμείτε παρακαλώ. Τώρα, λέει ο εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσα να εκφωνήσω ένα λόγο και να μείνω εδώ επί ώρε ασχολούμενο με το θέμα. Δεν το κάνω. Θα αναφερθώ σε κάποια σημεία τα οποία προαναφέρθηκαν. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά την κυρία Τσίμπερ, είπατε και δόθηκε η εντύπωση ότι υπήρξαν λέει, πολλές προσπάθειες να περάσει αυτή η οδηγία και φαίνεται ότι δεν τα καταφέρναμε και ότι όλο προβλήματα είχαμε μπροστά μας. Αυτό που, έχουμε, που είχαμε είναι ότι είμαστε στον τρίτο πυλώνα και έπρεπε να υποβληθεί μια πρόταση για απόφαση πλαίσιο. πλαίσιο. Και οι συζητήσεις προχωρούσαν καλά. Η απόφαση πλαισίου έπρεπε όμως να αποσυρθεί διότι έπαψε να ισχύει ο τρίτος πυλώνας και έπρεπε να υπανυποβάλουμε πρόταση σύμφωνα με τη νέα αρχιτεκτονική θεσμική δομή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι όλη η ιστορία για το τι συνέβη. Η πρόταση υποβλήθηκε το το Φεβρουάριο Φέτο. Συζητείτε τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα το περίεργο ή βραδύ ή αργό για το πώς προχώρησαν τα πράγματα πέρα από το γεγονός ότι η συνθήκη άλλαξε και οι πυλώνε άλλαξαν. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πέρα από το δικό μας έλεγχο και επιρροή και μπορούμε να πούμε ότι και μπορούμε να θεωρήσουμε θετικό αυτό το οποίο συνέβη. Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία περιγράφονται στην οδηγία. Εσείς ρωτήσατε όμως ποιος είναι αυτός που θα έχει πρόσβαση, ποιος θα συλλέγει, ποιος θα επεξεργάζεται αυτά τα δεδομένα και θα έχει πρόσβαση σε αυτά. Σας ε, αναφέρω στην ίδια την οδηγία. Λέτε ότι το φάσμα δεν θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευρύ και δεν θα πρέπει να περιορίζεται σε μικρά αδικήματα ή παραπτώματα. Όχι, περιορίζεται μόνο σε σημαντικά αδικήματα και παραπτώματα. Λέμε με σαφήνεια ότι πρέπει να υπάρχει μια ποινή που επισύρει ποινή τουλάχιστον τριετούς ε, φυλάκισης ώστε να μπορεί να δικαιολογείται η συλλογή και επεξεργασία στοιχείων. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί το επιχείρημα ότι για μικρά δικήματα και παραπτώματα αφορά, ασχολείται αυτή η οδηγία. Όχι, σας διασφαλίσω ότι δεν γίνεται αυτό. Μόνο σοβαρά δικήματα, εγκλήματα αφορώνται. Τώρα, στη συνέχεια, για την κυρία Ιντφέλτ, σε αυτά που είπε. Ένα γενικότερο σημείο το οποίο όμως πρέπει εδώ πρώτα να αναφέρω και αυτό είναι ότι η οδηγία, η οδηγία προβλέπει για την επιβολή του νόμου από τις αστυνομικές και διοκτικές αρχές να γίνεται ευφυής χρήση πολλών τεράστιων, ε, τεράστιου πλήθους στοιχείων και δεδομένων σε σχέση με την συμπεριφορά και στάση ενός υπόπτου. Αλλά αυτή η οδηγία, σε αυτή την οδηγία δεν υπάρχει αυτόματη διασύνδεση μεταξύ αυτόματου δεδομένου και επιπτώσεων όσον αφορά την επιβολή καταστολή. Πρέπει να υπάρχει ένα ανθρώπινο μυαλό, ένας άνθρωπος που να έχει μεσολαβήσει μεταξύ των δεδομένων, μεταξύ ανάλυσης δεδομένων και στοιχείων και την μετάφρασή τους σε λειτουργική δράση, η δίωξη. Δηλαδή πρέπει να υπάρξει παρέμβαση κάποιου ανθρώπου, κάποιου εγκεφάλου στο χτένισμα, στο κοσκίνισμα από αυτών των στοιχείων για την κατάληξη σε συμπεράσματα του τι πρέπει να γίνει σαν συμπέρασμα διανοητικά για αυτή την ε, κατάσταση. Και επίσης ε, κάτι άλλο πρέπει να δούμε εδώ. Το ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή οργάνωσε επίσης μαζί σας από κοινού και σε όλους σας που ενδιαφερόσαστε και πολλοί από σας ενδιαφερθήκατε και είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση μαζί σας που ενδιαφερόσαστε για τις αποδείξεις που είναι τεκμήρια και δείχνουν ότι το PNR ήταν απαραίτητο μέσο σε πολλές περιπτώσεις για την επίλυση πολλών εγκληματικών ερευνών και να κλειστούν στη φυλακή και να προσαθούν στη δικαιοσύνη και φυλακιστούν οι υπεύθυνοι εγκληματίε. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ήταν στοιχείο κλειδί το PNR για να φυλακιστούν αυτοί οι εγκληματίε. όταν υπήρχαν λόγοι και τεκμήρια που έπρεπε να μα ε, οδηγήσουν σε αυτή τη δράση. Αυτό που δεν μπορεί να επιλύσει αυτή η οδηγία και κανεί δεν μπορεί να επιλύσει και είναι θέμα πολιτική κρίση, είναι πόσε από αυτέ τι περιπτώσει είναι αναγκαίε για να διασφαλιστεί και να δικαιωθεί δικαιολογηθεί η ύπαρξη του συνολικού αυτού συστήματος. Και ο κύριος Χάστινγκς ο ίδιος, ο επικεφαλής ε, της μονάδας, μου είπε εμένα και είπε και σε εσά σε μια ακρόαση για την αποθήκευση στοιχείων προσωπικών δεδομένων ότι είναι αυτό μια αξιολόγηση, μια κρίση που μόνο πολιτικά μπορεί να ληφθεί ως απόφαση. Μετά όμως από τα στοιχεία τα οποία έχουμε και σας δώσαμε είναι απαραίτητο και είναι σαφές ότι είναι απαραίτητο το PNR για την δίωξη των εγκλημάτων εγκληματιών. Θα ήταν ανεύθυνο από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αγνοήσουμε τη σπουδαιότητα αυτών των τεκμηρίων που μα δόθηκαν από τι διοκτικέ αρχέ των κρατών μελών και να μην δίναμε συνέχεια και να μην υποβάλαμε αυτή την πρόταση προς έγκριση σε εσά. Ο κύριος Ευρωβουλευτής Άλμπρεχτ έθιξε το ζήτημα της ανωνυμίας. Μπορώ να σας διασφαλίσω ότι σύμφωνα με την ίδια την οδηγία τα στοιχεία αυτά θα είναι ανώνυμα μετά από ένα μήνα ήδη κιόλα στην αποθήκευσή τους. Θα έχουν αποπροσωποιηθεί, δεν θα είναι δηλαδή ονομαστικά δεσμευτικά για κάποιον, δεν θα χαρακτηρίζουν κάποιον πλέον. από πλευράς ε, ε, Ευρωβουλευτού Έρνστ τέθηκε το θέμα αν η οδηγία για τα προσωπικά δεδομένα δεν θα έπρεπε να εγκριθεί πριν από αυτή την οδηγία εδώ νομίζω υπάρχει κάποια παρανόηση πρέπει να σας πω. Χρειάζεται ένας γενικότερος νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων φυσικά. Υπάρχουν οι γενικές αρχές για την προστασία των ε, προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τη χάρτα και τα συντάγματα. Μετά χρειάζεται ένα γενικό νομικό πλαίσιο, ένας γενικός νόμος λέγοντας ποιε είναι οι γενικές αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων και μετά κάθε σύστημα για την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα θέλει, απαιτεί ειδικού εξειδικευμένους νόμους και κανόνες για την πρόσβαση. Αν θέλετε να έχουμε σημαντικές δικλείδες και προδιαγραφές για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σε αυτή την πρόταση, πράγμα που καλωσορίζουμε, πρέπει να υπάρξει ένα σύστημα προστασίας προσωπικών δεδομένων σε αυτό το σύστημα, άσχετα από ποιοι κανόνες υπάρχουν στο γενικό μέσο ή σε γενικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων. Λαθασμένη συζήτηση ήταν, θα ήταν να λέγαμε πρώτα να υπάρξει μια οδηγία για την προστασία, στο μέλλον βέβαια, για την προστασία προσωπικών δεδομένων προτού ρυθμίσουμε και εγκρίνουμε αυτή την πρόταση και μετά να συνεχίσουμε. Λάθος θα ήταν αυτό. Μετά στη συνέχεια υπάρχει κάτι άλλο για το, την παρέμβαση της κυρίας Λάντφορντ. Για άγνωστους λέει υπόπτους. Αυτή η οδηγία δεν μετατρέπει, δεν μεταθέτει άτομα, ανθρώπους, δεν τους κάνει εγκληματίες. Είναι τα εγκλήματά τους που τους κάνουν εγκληματίες. Αυτή η οδηγία απλά διευκολύνει, διευκολύνει την ζωή των διοκτικών αρχών και των δικαστικών αρχών στο να καταδείξουν και να αποδείξουν με τεκμήρια το ότι κάποιοι έχουν εγκληματίσει στο παρελθόν και έχουν διαπράξει εγκλήματα. Αυτό δεν δημιουργεί περισσότερους υπόπτους ή περισσότερους εγκληματίες, απλώς διακριβώνει ποιοι είναι οι εγκληματίες που αλλιώς δεν τους βρίσκαμε. Όλοι συμφωνούμε ότι εκείνοι που έχουν διαπράξει εγκλήματα θα πρέπει, θα έπρεπε να προσαχθούν στη δικαιοσύνη και να καταστούν ε, να υπομισθούν τις ευθύνες των πράξεών τους και να δικαστούν με βάση αυτές και καταδικαστούν και σε σχέση με την αποπροσωποποίηση των προσωπικών δεδομένων μετά από περίοδο ενό μήνα. Πράγματι, θεσπίσαμε ότι μετά από ένα μήνα η ταυτότητα του ατόμου που, από το οποίο έχουν συλλεγεί αυτά τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι προσπελάσιμη στις αρχές εκτός αν πάρα πολύ σημαντικοί λόγοι θα οδηγούσαν θα οδηγούσαν τις διοκτικέ αρχές ή του δικαστές στο να έχουν τελικά πρόσβαση σε αυτό το όνομα και αυτά τα στοιχεία σε σχέση με τεκμηριωμένες υποψίες. Αλλά η, τα, τα στοιχεία αυτά δεν θα ήταν πλέον διαθέσιμα για ανάλυση ή επεξεργασία ή ένα είδο συμπεριφοράς. Αυτά θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή. Ευχαριστώ. Ελπίζω να μην χρονοβόρησα, να μην μακρηγόρησα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια που κάνατε να μας εξηγήσετε τη φύση και το περιεχόμενο της ε, οδηγίας ε, που προτάθηκε. Τώρα θα ήθελα να στραφώ και πάλι προς τον εισηγητή μας, τον κύριο Κίρκοπ, για να συνοψίσει τέλος πάντων αυτό το πρώτο στάδιο ε, της πρωτης ανταλλαγής απόψεων 1α όπως τη χαρακτήρισαμε προηγουμένω. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα τα σχόλια που άκουσα. Θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα-δυο. Σε σχέση με τα σχόλια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καταρχάς, είναι πάρα πολύ σημαντικά και συμφωνώ με ε, τον συνάδελφο σε πολλά σημεία, όμως ε, οι προτάσεις ε, της Επιτροπής είναι το σημείο αφετηρίας και όχι το τέλος της διαδικασίας αυτής. Άκουσα λοιπόν αυτά που είπε. Η δική μου έκθεση ελπίζω να έχει τα δικά της χαρακτηριστικά, διαφορετικά από την πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα τα συζητήσουμε βέβαια και στο πλαίσιο της Επιτροπής μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όσον αφορά τα σχόλια του, Συμβουλίου, συγγνώμη, ναι, πράγματι μας ενδιαφέρει σε τελική ανάλυση η κατάχρηση των ενδιαφερομένων μερών. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν εμφανιστεί ως τέτοιοι ακόμα και βεβαίω θέλουμε να λάβουμε υπόψη αυτά τα οποία θα πούν, όμω στο τέλο τη διαδικασία, ένα μόνο κείμενο υπάρχει. Και το κείμενο δεν, μπορεί, δεν μπορούμε να έχουμε 100 κείμενα που να αντικατοπτρίζουν τι απόψει όλων των ενδιαφερομένων για όλα τα πράγματα. Για τη Σοφή Νετφελτ λυπάμαι που έπρεπε να φύγει, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνόμαστε με την ε, κυρία Ινετφελτ ε, και αυτό φανήκε και σε άλλα ζητήματα που έχουμε συζητήσει, σε παρόμοια παρόμοιους τομείς. Ε, τα θέματα που αφορούν τα δεδομένα και που έθεσε είναι πράγματι ανησυχητικά. Η αποθήκευση των δεδομένων, από ποιον, πού, για πόσο χρονικό διάστημα, ε, ο χαρακτηρισμός των δεδομένων, η φύση τους, η χρήση των βάση, της δεδομένων, ε, ε, τη χρήση των δεδομένων αυτών. Χρειαζόμαστε πολύ σαφείς και αυτό είναι κάτι στο οποίο θέλουμε να στρέψουμε σύντομα την προσοχή μας. Και η κυρία Χέντς και ο κύριος Άλμπρεχτ έχουν ε, επιφυλάξεις. Όλες οι μεγάλες πολιτικές ομάδες μίλησαν σήμερα εκτός από μία. Υπάρχουν επιφυλάξεις, καταλαβαίνω απολύτως επιφυλάξεις αυτές. Ε, ελπίζω να μπορέσω να ικανοποιήσω τον κύριο Άλμπρεχτ και την κυρία ε, ε, Χέρς ανάλογα Βέβαια με το τι ακριβώς θα ζητήσουν θα ήθελα να πω προς τον κύριο Άλμπρεχτ ότι οι νομικές γνωμοδοτήσεις είναι εξίσου σημαντικές με τις υπόλοιπες, είναι όμως γνωμοδοτήσεις. Νομίζω ότι το είπα και προηγουμένως. Η κυρία Χέρς δεν συμφωνεί νομίζω με τη συμφωνία PNR, τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Ε, δεν μπορώ, ελπίζω να μπορέσω να, τις, να την πείσω κάπως ότι έχει νόημα αυτή η συμφωνία. Όσον αφορά τώρα τη χρήση, τη χρησιμότητα μάλλον ε, της PNR. Κάτι κατά πόσο υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι χρησιμοποιήθηκε το PNR για την ε, σύλληψη την παρεμπόδιση, τη σύλληψη τρομοκρατών ή την παρεμπόδιση τρομοκρατικών πράξεων. Όλοι όσοι μπορέσατε να αποδεχτείτε την πρόσκλησή μου στο Μάντσεστερ ε, θα είδατε ε, κάποια από τα αποδεκτικά αυτά στοιχεία και κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας ελπίζω να μπορέσουμε να ε, βρούμε και άλλου τέτοιου είδους παρατήρηση και άλλου τέτοιου παραδείγματα, συγγνώμη. Τώρα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ναι, είναι πολύ σημαντικό ε, τα ανθρώπινα δικαιώματα των ανθρώπων όμως που μπορεί να χάσουν τη ζωή τους λόγω τρομοκρατικής ε, πράξης είναι κάτι το οποίο εμένα με απασχολεί πάρα πολύ. Ε, ο, το είδος των αδικημάτων που θα αφορά βέβαια το θέμα αυτό Συγγνώμη, ελπίζω να μην φταίω εγώ που πέσατε. Okay, I oh, Α, τότε εντάξει, είστε καλά. Ε, εν πάση περιπτώσει τη φύση των αδικημάτων πρέπει να την ε, ε, προσέξουμε όντως άλλο είναι μια ποινή τριετούς φυλάκισης άλλο είναι άλλα πράγματα θα ήθελα να δω ορισμούς πολύ συγκεκριμένους σαφέστερους για να βλέπουμε να είναι σαφές ότι μιλάμε ειδικότερα για σοβαρά δικήματα και τρομοκρατία τώρα το θέμα του profiling το οποίο το έθεσε η Βαρόνι Λάτφορντ νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Πρέπει να προσμετρήσουμε τα στοιχεία αυτά, γιατί η έμεση διάκριση είναι ένας πολύ ευρύς τομέας. Ε, οι διακρίσεις μπορεί να είναι έμεσες ε, ε, και μάλιστα να γίνονται με τρόπο που πολύ συχνά δεν τον σκεφτόμαστε και πρέπει να μας απασχολήσει και αυτό. Επίσης, ανέφερε η Βαρόνι Λάντφορτ ε, αν υπάρχει ένα πλαίσιο το οποίο εκπληρώνει το σκοπό μας ή κάπως έτσι το είπατε. Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι αυτό το πλαίσιο είναι το πλαίσιο PNR και ότι μπορούμε να ε, βασιστούμε στα στοιχεία που περιλαμβάνει το πλαίσιο αυτό για να μπορέσουν να προστατευτούν τα προσωπικά δεδομένα των ανθρώπων. Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Κίρκοπ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σημαντική συζήτηση αυτή καλή χορταστική για την πρώτη α φάση 1A για αυτή τη φάση διαπραγμάτευσης. Δεν έχουμε φτάσει στην 1β ακόμα, αλλά σχεδόν. Και θα έλεγα ότι Συνεχίζουμε και είμαστε έτοιμοι να δώσουμε συνέχεια αμέσως μετά τις ε, θερινές διακοπές, με τα επόμενα βήματα που θα κάνουμε και πρέπει να γίνουν στο πρόγραμμα εργασίας της δικής μας Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, δίνοντας συνέχεια σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό χαρτοφυλάκιο στις εργασίες μας. Προτείνω να συνεχίσουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη. Συνεχίζουμε και πάμε στο σημείο 20. Μάλιστα. Σημείο 20. Αυτό αφορά ένα μηχανισμό αξιολόγησης για την επαλήθευση και εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγγεν. Πολύ καλά. Λοιπόν, αν είσαστε αρκετά ευγενικοί να εγκαταλείψετε την αίθουσα ήσυχα εκείνοι οι οποίοι θέλετε να αποχωρήσετε ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε με τη δουλειά μας εμείς που θα παραμείνουμε. Μάλιστα.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 colleagues, we are here to keep on with our work. Να συνεχίσουμε λοιπόν συνάδελφοι, εντάξει. Deal now. Πολύ καλά. Λοιπόν θα εξετάσουμε τώρα την παρουσίαση τη γνωμοδότηση των νομικών υπηρεσιών, τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα παρουσιάσει η νομική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου την άποψή τη, την γνωμοδότησή τη για τη νομική βάση όσον αφορά την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αξιολόγηση του κεκτημένου του Σέγγεν. Ξέρουμε ότι ο κύριος εισηγητής είναι ο κύριος Κουέλιο που υπέβαλε το σχέδιο έκθεσης του στις 2 Μαΐου. Η δική μας Επιτροπή ΛΥΜΠΕ έκανε συζήτηση για τις τροπολογίες στις 16 Ιουνίου και ο εκπρόσωπος της Προεδρίας ενημέρωσε ότι σταμάτησε τις εργασίες του επί της ουσίας αυτής της πρότασης στο Συμβούλιο. Με βάση μια γνωμοδότηση λοιπόν των νομικών υπηρεσιών του Συμβουλίου που εξετάζουν την αλλαγή της νομικής βάσης στο άρθρο 70 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η νομική βάση που επελέγει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή άρθρο 77 2 ε της Συνθήκης Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπει τη διαδικασία συναπόφασης ενώ το άρθρο 70 δεν προβλέπει καμιά εμπλοκή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην νομοθετική διαδικασία, στο νομοθετικό έργο. Σαν συνέπεια λοιπόν δικού μας αιτήματο, αιτήματο του εισηγητή, ζήτησα ως πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, ΛΥΜΠΕ, από την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συντάξει μια γνωμοδότηση για το τι γίνεται σε σχέση με την, το εύθετο της νομικής βάσης αν μπορεί να γίνει δεκτή ή όχι. Επίσης ζήτησα να εξετάσει η νομική μας υπηρεσία σε ποιο βαθμό το ευρώ τη πρόταση μπορεί να διευρυνθεί ώστε να καλύπτεται η καταπολέμηση της διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματος επίσης. Μια και αυτό είχε ζητηθεί με διάφορες τροπολογίες ω αίτημα. Τώρα θα ακούσουμε την παρουσίαση της ε, νομικής αυτής γνωμοδότησης ε, που συντάχθηκε από τη νομική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου. Στη συνέχεια θα ακούσουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα σχολιάσει και μετά θα έχουμε τα σχόλια της Προεδρίας του Συμβουλίου και μετά έχοντας ακούσει και τον εισηγητή μας κύριο Κουέλιο και άλλα μέλη θα συνεχίσουμε. Έτσι λοιπόν ο εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας είναι η κυρία Ντίν από ό,τι γνωρίζω. Μπορείτε να παρουσιάσετε τη νομική γνωμοδότηση παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Thank Σας ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτή την ευκαιρία να παρουσιάσουμε την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας για μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα κανονισμό για τη θέσπιση ενός μηχανισμού αξιολόγησης για την επαλήθευση της εφαρμογής του κεκτημένου του Σέγγεν. Στην επιστολή σας θέτετε τέσσερα ερωτήματα. Πρώτον, για τη σωστή νομική βάση. Δεύτερον, τις επιπτώσεις σε σχέση με την επιλογή του άρθρου 70 ως νομικής βάσης. Τρίτον, τη δυνατότητα να συνδυαστούν τα άρθρα 77 με το άρθρο 70, τα δύο άρθρα 77 και 70 Τέταρτον, τη δυνατότητα διεύρυνσης του νομικού φάσματος και για άλλες χρήσεις. Λοιπόν, για την νομική βάση που προτείνεται την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, <clears throat> άρθρο 70 ε, που προβλέπει μέτρα σε σχέση με ελέγχου ε, όσον αφορά άτομα που διασχίζουν τα εσωτερικά σύνορα η αιτιολογία είναι ότι η κατάργηση των ελέγχων των εσωτερικών συνόρων, που είναι ο τελικό στόχο σε σχέση με την ελευθερία τη κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, συμφωνούμε με αυτή την ε, επεξήγηση. Θεωρούμε όμω ότι το άρθρο 70 ε, ε αυτού δεν επαρκεί ως νομική βάση αυτό μόνο του ο ενιαίος χώρος για την ελευθερία κυκλοφορίας των ατόμων και για την κατάργηση των ελέγχων στα σύνορα η κατάργηση των εσωτερικών ελέγχων στα σύνορα απαιτεί την εφαρμογή ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα ως προϋπόθεση. Είναι οι δύο όψεις ενός νομίσματος και κοινοί κανόνες απαιτούνται για να εφαρμοστούν όλα αυτά. Κοινοί κανόνες κοινοτικοί κανόνε και κανονισμοί σε σχέση με του ελέγχου στα εξωτερικά σύνορα και την ελευθερία κυκλοφορία των ατόμων. Το άρθρο 77.1 λέει και προβλέπει ότι ο στόχο είναι οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα. Πρέπει να βελτιωθούν οι έλεγχοι στα εξωτερικά σύνορα. Το 77.2 προβλέπει και δίνει τη νομική βάση για την υιοθέτηση και έγκριση των αναγκαίων μέτρων. Γι' αυτό εμεί θεωρούμε στη γνωμοδότησή μα ότι η σωστή βάση είναι ω επιλογή το άρθρο 77 παράγραφο 2 σύνολο Επιπρόσθετα, θεωρούμε ότι το άρθρο 74 θα πρέπει και αυτό να προσθεθεί στη νομική βάση που θα επιλεγεί ώστε στην πρόταση αυτή να υπάρχουν υποχρεώσει από τα κράτη-μέλη να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο έργο αυτό. Η προσθήκη του άρθρου 74 δεν θα είχε επιπτώσει στην εφαρμογή τη κανονική νομική νομοθετικής διαδικασίας στη συναπόφαση. Σε σχέση λοιπόν με το πρώτο ερώτημα, η σωστή νομική βάση είναι το άρθρο 77 παράγραφος 2 και το άρθρο 74 τη συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Περνώντα στο δεύτερο ερώτημά σα μας ρωτήσατε και ζητήσατε ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις της χρήσης του άρθρου 70 ως νομικής βάσης. Επιπρόσθετα στο γεγονός ότι ο ρόλος του Ευρωκοινοβουλίου θα άλλαζε υπό το άρθρο 70 το Ευρωκοινοβούλιο απλώς θα ενημερωνόταν, δεν θα συναποφάσιζε. Το άρθρο 70 προβλέπει ότι το Συμβούλιο μπορεί να καθορίσει ρυθμίσει και διατάξει σύμφωνα με τι οποίε τα κράτη-μέλη σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγουν αντικειμενικέ και αμερόληπτες αξιολογήσεις σε σχέση με τα μέτρα που ε, υιοθετούνται από τα κράτη-μέλη. Δηλαδή τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που είναι αρμόδια για την αξιολόγηση της εφαρμογής από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Είναι ένα σύστημα για αμοιβαία αξιολόγηση και αποτίμηση από τα ίδια τα κράτη-μέλη. Η εξουσία για την άσκηση αυτής της ε, αξιολόγησης είναι των κρατών μελών και έτσι εμείς πιστεύουμε ότι το άρθρο 70 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νομική βάση για να υπάρξει η δημιουργία ενός μηχανισμού αξιολόγησης ε, <clears throat> όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αρμόδια για την εφαρμογή αυτών των ε, διατάξεων αξιολόγηση, όπου θα είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδια για την ε, αξιολόγηση αυτών που έχουν ε, γίνει από τα κράτη-μέλη. Επιπλέον το άρθρο 70 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν οι συστάσει θα έχουν επιπτώσει στο κεκτημένο του Σέγγεν. Όπως θα συνέβαινε αν υπήρχαν υποχρεώσεις όσον αφορά κυρώσει όσον αφορά τα κράτη-μέλη. Το τρίτο ερώτημα που διατυπώσατε, αν θα ήταν δυνατόν να συνδυαστούν τα άρθρα 77 και 70. Εμείς θεωρούμε ότι δεν θα ήταν δυνατόν να προσθεθεί στην στη νομική βάση τη σημερινή πρόταση του άρθρου 70. Στη σημερινή πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρμόδια για την αξιολόγηση και εφαρμογή του μηχανισμού αξιολόγηση. Τέταρτο ερώτημα που διατυπώσατε. Αν το εύρο, το φάσμα των έργων των αρμοδιοτήτων θα μπορούσε να διευρυνθεί για την καταπολέμηση τη διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματο. Πρώτον, η καταπολέμηση τη διαφθορά και του οργανωμένου εγκλήματο δεν είναι μεταξύ των στόχων του κεκτημένου του Σέγγεν. Και δεύτερον, ο στόχος του μηχανισμού αξιολόγησης είναι η αξιολόγηση της, εφάρμοσης, της εφαρμογής του ΑΚΙ και όχι η ερμηνεία, η θέσπιση νέων διατάξεων. Ωστόσο, η καταπολέμηση της διαφθοράς και της, του οργανωμένου εγκλήματος και που μας κάνει να δούμε την, ανεπαρκή, την ανεπάρκεια της εφαρμογής του κεκτημένου του Σέγγεν και αυτό το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπονόμευση είναι κέρια σημασία για την αξιολόγηση. Ευχαριστώ για την προσοχή. Και εμείς σας ευχαριστούμε και ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Τώρα να ακούσουμε τον εισηγητή μα τον κύριο Κοέλη. so much, Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω την νομική υπηρεσία για την ταχεία αντίδρασή της ε, στο αίτημά μας ε, που ε, έγινε στην τελευταία μα συνεδρίαση όπω είπε ήδη ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία ζητήματα. Στη νομική βάση, στη διαφθορά ε, και στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία. Σε σχέση με, το, με τη νομική βάση θα ήθελα να ευχαριστήσω ε, για, την, ε, για τις συμβουλές της στη νομική υπηρεσία και χαίρομαι ιδιαιτέρως που διαπιστώνω ότι υποστηρίζει την προσέγγιση η νομική υπηρεσία υποστηρίζει την δική μου προσέγγιση που εμφανίζεται και στην έκθεσή μου αλλά και την προσέγγιση της Επιτροπής μας. Θα ήθελα να τονίσω αυτό που μόλις είπε η νομική υπηρεσία. Το άρθρο 70 δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για ε, την απόδοση ε, ε, εφαρμοστικών εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οτιδήποτε αναφέρεται στο άρθρο 70 δεν μπορεί να επηρεάσει, δηλαδή για τις νομοθετικές πράξεις δεν μπορεί να επηρεάσει το κεκτημένο του Σέγγεν όσο έχει αυτή τη στιγμή ούτε να επιβάλλει την υποχρέωση στα κράτη-μέλη να οδηγήσει σε κυρώσεις. Επομένως, οποιαδήποτε απόφαση που ε, λαμβάνεται υπό το άρθρο 70 θα αποτελούσε ε, μόνο ε, τμήμα του τρέχοντος μηχανισμού αξιολόγησης της Έγγεν. Τι συμβαίνει τώρα. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην τελευταία του συνεδρίαση αποφάσισε και παραθέτω Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν κενά ε, στο, και και εκτιμένο της έγκαινο όσον αφορά την ε, πραγματική εφαρμογή και την επιβολή της ισχύουσας νομοθεσίας. Και επίσης το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αναφέρει ότι η ενίσχυση ε, του μηχανισμού αξιολόγησης του Σέγγεν που πρέπει να αποτελέσει ένα μηχανισμό αποτελεσματικότερο για την καλύτερη εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγγεν και καλύτερη θεσμική ισορροπία μεταξύ κρατών μελών ε, και ευρωπαϊκών θεσμών θα έπρεπε να εξεταστεί. Αυτό ε, σημαίνει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν βλέπει, δεν εξετάζει το πρόβλημα αυτό μόνο για την αξιολόγηση του κεκτημένου του Σέγγεν, αλλά ζητούν την αλλαγή των ε, νομικών μέσων ε, που αφορούν τον μηχανισμό αξιολόγησης. Άρα, το άρθρο 70 δεν μπορεί να αποτελέσει τη νομική βάση. Και σε προηγούμενη συνεδρίαση είχα πει ότι το γεγονός ότι ζήτησαν την αλλαγή της νομικής βάσης πολλά κράτη-μέλη ε, ήταν ε, μια πολιτική εχθρική πράξη εναντίον του Κοινοβουλίου. Ήταν ε, μια λανθασμένη κίνηση όταν ζητούμε την καλύτερη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ήταν όμως μόνο μια εσφαλμένη πολιτική κίνηση τελικά είναι και ανοησία. Γιατί με αυτή τη νομική βάση ο στόχος, ο πολιτικός ε, ε στόχος, εν πάση περιπτώσει, ε, που ζήτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δεν μπορεί να εκπληρωθεί. Οπότε, Ευχαριστώ όλος ιδιαίτερος ε, τη νομική υπηρεσία για τη γνωμοδότησή της. Για μένα είναι σαφές ότι δεν μπορούμε να επιτύχουμε τις αλλαγές που θέλουμε με το άρθρο 70. Το άρθρο 77 σε συνδυασμό με το άρθρο 74 όπως ε, πρότεινε και η νομική υπηρεσία θα έπρεπε να αποτελούν τη νομική βάση και ε, θα έπρεπε να ε, κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να θέσω, η διαφθορά. Η γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας, ε, της νομικής υπηρεσίας μας επιβεβαιώνει αυτά που είπα την προηγούμενη, στην προηγούμενη συνεδρίαση. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε την, το κεκτημένο του Σέγγεν μέσω αυτής της πρότασης. Η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς δεν ε, είναι μεταξύ των στόχων ε, της, του κεκτημένου του Σέγγεν ο σκοπός του μηχανισμού είναι να επιβεβαιώνει την εφαρμογή του κεκτημένου του Σέγγεν και όχι να ορίζει νέα κριτήρια. Όμως, ε, επειδή οι στόχοι του κεκτημένου του Σέγγεν συμπεριλαμβάνουν τη βελτίωση της αστυνομική και της δικαστικής συνεργασία σε ποινικά ζητήματα, θα μπορούσαμε να συμπεριλάβουμε σε αυτόν τον μηχανισμό μια αξιολόγηση του κατά πόσο ε, ε, υπάρχουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με την αποτυχία των κρατών μέλων αντιμετώπισης ε, της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος που αποδυναμώνουν, δημιουργούν πρόβλημα στην εφαρμογή ε, του κεκτημένου της Schengen. Οπότε νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συντάξουμε μια συμβιβαστική πρόταση ε, υπ' αυτήν την έννοια. Και το τελευταίο θέμα, κύριε Πρόεδρε, που θα ήθελα να θέσω σε σχέση με την ε, κατάσταση της Ιρλανδίας και του Ηνωμένου Βασιλείου. Εγώ παρουσίασα κάποιες ε, τροπολογίες, όπως και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το ζήτημα που, έχει, να, που αφορά ε, την συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας στον τρίτο πυλώνα, που σκοπό έχει να δίνει τη δυνατότητα στι χώρε αυτέ ε, να αξιολογούν ε, στο πλαίσιο της αστυνομικής συνεργασίας ε, ε, το, την παροχή σχετικών δεδομένων. Η άποψη λοιπόν της νομικής υπηρεσίας μας λέει ότι θα ήταν καλύτερο να υπάρξει ένα ξεχωριστό μέσο για τη συμμετοχή αυτή. Ε, θα ήθελα να ρωτήσω την νομική υπηρεσία αν κατά την άποψή της η πρόταση, η λύση που προτείνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την ε, Ιρλανδία και το Ενωμένο Βασίλειο στο πλαίσιο ε, της υπηρεσίας ε, αυτής θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στην επόμενη πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρος, και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ήταν ε, πολύ σαφής η παρουσίαση της άποψή σας και υπάρχει έτοιμα να συζητηθεί. Βλέπω μέλη που ζήτησαν τον λόγο, αλλά πρώτα θα ακούσουμε την Επιτροπή. Κυρία Μόσχαμερ, παρακαλώ. Μόσχαμερ, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τη νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή τη γνωμοδότηση που έδωσε. Δυστυχώ την πήραμε μόνο πολύ πρόσφατα με καθυστέρηση και θα σχολιάσω μόνο το κύριο τμήμα, το πιο σημαντικό τμήμα. Θέλω παρόλα αυτά να εκφράσω υποστήριξη για το άρθρο 77 ως νομική βάση, όπως το είχε ταυτοποιήσει, εντοπίσει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης και για την προσθήκη στη συνέχεια του 74 φυσικά θα αναλύσουμε κατά λεπτό τα επιχειρήματά σας από πλευράς μας. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν να βελτιωθεί ο σημερινός μηχανισμός. Όλοι συμφωνήσαμε, συμφωνούμε ότι έχει κενά χάσματα, ε, ευάλωτα σημεία αυτή η σημερινή κατάσταση και έπρεπε να βελτιωθεί. Και ο κύριος Κοέλιο το είπε και το Συμβούλιο ότι πρέπει να βελτιωθεί η αξιολόγηση, ο μηχανισμός αξιολόγησης του Σέγγεν. Πρέπει να υπάρχει ένας ενδυναμωμένος μηχανισμός και σε αυτή τη γραμμή, όπως τόνισε και η νομική υπηρεσία, υπάρχει ανάγκη να επανορθωθούν αυτές οι αδυναμίες και πρέπει αυτό να είναι σαφές και πρέπει να υπάρχουν και κυρώσεις κατά κάποιο μέτρο για να επανορθωθούν, να βελτιωθούν οι αδυναμίες που έχουν εντοπιστεί σε σχέση με τη σωστή ορθή εφαρμογή του κεκτημένου και εν τέλει τη λειτουργία της περιοχής της ζώνης Σέγγεν ως σύνολο ω συνόλου. Και γι' αυτό είμαι ευγνώμων για το ότι οι νομικές υπηρεσίες υποστήριξαν την επιλογή της νομικής βάσης με αυτόν τον τρόπο. Όσον αφορά τη διεύρυνση του φάσματος όσον αφορά το κεκτημένο για την καταπολέμηση τη διαφθορά. συμφωνώ ότι η διαφθορά και η καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος μέρος τη αξιολόγησης εφαρμόζοντας το κεκτημένο και όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία θα πρέπει αυτό υστερότερα να το εξετάσουμε. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για το Συμβούλιο. Πολωνική Προεδρία. Ο κύριος Μπογκουντέτσκι παρακαλώ. Το πρόφερα σωστά. Έχετε τον, τον λόγο αν επιθυμείτε παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Καλό σας απόγευμα. Λέγομαι, λέγομαι Μπογιουσέσκι. εργάζομαι στο Συμβούλιο όπου εκπροσωπώ και την Δημοκρατία της Πολωνίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχω την τιμή να εκπροσωπώ εδώ την Πολωνική Προεδρία κατά τις συνεδριάσεις με την Επιτροπή σας. Λαμβάνοντας υπόψη τις δηλώσεις του Υπουργού μου σε αυτή την αίθουσα πρέπει να σας πω ότι η προτεραιότητα της Πολωνικής Προεδρίας είναι να συνεργαστεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα πλαίσια αυτών των θεματικών. Και πρέπει να, το, να παρακολουθήσουμε όλα αυτά τα θέματα όσο το δυνατόν πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Κατά βάθος η Προεδρία θεωρεί ότι το πρόβλημα το οποίο εξετάζετε εσείς έχει και κάθετο και οριζόντιο χαρακτήρα. Μιλάμε για τη νομική βάση η οποία να καλύπτει την πρώτη και τη δεύτερη φάση της εντολής αξιολόγησης του Σέγγεν και να εγγυάται και την εμπλοκή σε όλη τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπως επίσης και αν χρειαστεί η επέκταση της πρότασης. η Πολωνία ως Προεδρία θέλει να αναζητήσει ένα συμβιβασμό στο Συμβούλιο για αυτά τα θέματα. οι βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ενημερωθούν για όλα όσα θα συμβαίνουν στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου. Εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να βρούμε ένα συμβιβασμό σε αυτή την ιστορία. Το Σεπτέμβριο φέτος θέλουμε να ολοκληρώνουμε. Τώρα για τις προθεσμίες να σας θυμίσω κυρίες και κύριοι ότι προετοιμάζεται μία συζήτηση στο ΣΟΠΟΤ στις 18 Ιουλίου. Ωραία. Θα ήταν χρήσιμο η νομική υπηρεσία να απαντήσει σε αυτά τα ε, συγκεκριμένα ερωτήματα που έθεσε και ο εισηγητής ο κύριος Κοέγιο ε, ο αίσθηση ο Κοέγιο. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κοέγιο μας ρώτησε κατά πόσο θα, ήταν, ε, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε την πρόταση που εφαρμόστηκε για την υπηρεσία IT. Σε σχέση όμω με αυτήν την υπηρεσία, το Ηνωμένο Βασίλειο είχε ζητήσει επί τη βάση του άρθρου 4 του πρωτοκόλου τη ΕΝΓΕ να συμμετέχει σε κάποιε διατάξει του κεκτημένου τη ΕΝΓΕ και αυτό ε, εγκρίθηκε από το Συμβούλιο με απόφαση του Συμβουλίου και το Ηνωμένο Βασίλειο μπόρεσε να συμμετέχει έχει πλήρως στην έγκριση του κανονισμού της συγκεκριμένη υπηρεσίας. Το αίτημα έγινε για να συμμορφωθούμε με την ομολογία του δικαστηρίου βάσει της οποία πρέπει να συμμετέχουμε ε, στο συγκεκριμένο τμήμα του κεκτημένου πριν συμμετέχουμε ε, σε ένα ε, μέτρο ε, που οδηγεί στην εφαρμογή αυτού του κεκτημένου. Το Συμβούλιο μπορούσε να, ακολουθήσει, να επιλέξει να ακολουθήσει την ίδια ε, προσέγγιση, όμως αυτή είναι μια διαδικασία η οποία επαφίεται απολύτως στο Συμβούλιο, δεν υπάρχει καμία συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν υπάρχει κανένα, καμιά υποχρέωση ενημέρωσης ή διαβούλευσης με το Κοινοβούλιο. Αν το Συμβούλιο επιλέξει να ακολουθήσει τη διαδικασία αυτή, θα επέτρεπε στο Ηνωμένο Βασίλειο να συμμετέχει πλήρως. Αλλά ελήψη τέτοιας απόφασης ε, δεν βλέπω πώς θα ήταν δυνατό. Κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να υπάρξουν δύο διαφορετικές προτάσεις. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Νεντέλτσεβα θέλει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ τους ομιλητές για όλη η όσα μας είπαν όπως και τη νομική υπηρεσία του Κοινοβουλίου που αποδεικνύει και τη συνέχεια της θέσης, τη λογική συνέχεια της θέσης που εμείς προασπιζόμαστε. Εμείς ε, σε αυτή τη γνωμοδότηση βλέπουμε τέσσερα σημεία. Η νομική υπηρεσία επιβεβαιώνει αυτό το οποίο είχαμε πει από την αρχή. 77 ε, παράγραφος 2 και 74. Αυτές είναι οι νομικές βάσεις. Είναι πολύ σημαντικό κάθε φορά να θυμόμαστε ότι αυτός ο μηχανισμός του Σέγγεν πρέπει να βασίζεται σε μια κοινοτική μέθοδο να σέβεται το κοινοτικό πνεύμα και αυτό με αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Δεν θα πρέπει να χειραγωγηθεί το Σέγγεν για την εξυπηρέτηση εθνικών ε, βράχυπρόθεσμων συμφερόντων. Πρέπει να προσπίσουμε το ρόλο του Κοινοβουλίου που, εκλέγεται άμεσα από τους πολίτες. Η περιθωριοποίηση του Κοινοβουλίου θα στείλει ένα μήνυμα ότι παραμερίζεται και ο πολίτης και δεν είναι κατάλληλη στιγμή να γίνει κάτι τέτοιο σήμερα με την κρίση που περνάμε. Επιπλέον, πώς θα ενισχύσουμε Τι θέση μας μετά τη συνθήκη της ε, Λισαβόνας που προβλέπει ότι με το Συμβούλιο θα πρέπει να συναποφασίζουμε. Όλοι έχουμε συνειδητοποιήσει ότι ο τωρινός μηχανισμός του Σέγγεν πρέπει να ενημερωθεί. Αυτό πρέπει να γίνει με ένα καθεστώς διαφάνειας για να έχει νομιμότητα. Και ο τωρινός ενημερωμένος μηχανισμός θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το ίδιο από όλα τα κράτη-μέλη χωρίς να επιφέρει σημαντικό γενικότερες επιβαρύνσεις για τη μία ή για την άλλη χώρα. Οπότε πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα στο Συμβούλιο ότι εμείς βασιζόμαστε σε αυτές τις αρχές, αυτές είναι οι αξίες μας και καλό θα ήταν και το Συμβούλιο να το, να το πράξει. Τώρα για την διαφορά. Συμφωνώ με αυτό το οποίο είπε ο κύριος Κοέγιο. Η καταπολέμηση της ε, διαφθοράς ε, δεν είναι εκτιμένο του Σέγγεν. Έχουμε πολλούς μηχανισμούς που ασχολούνται με αυτό και δεν μιλάω για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία που έχουμε το μηχανισμό επαλήθευσης της ε, συνεργασίας. Αλλά στις αρχές Ιουνίου η κυρία Μάλστρομ μας παρουσίασε τη στρατηγική της κατά της διαφθοράς. Είναι το πιο φιλόδοξο έγγραφο το οποίο είδαμε τα τελευταία χρόνια και αν θέλουμε να είμαστε πιστικοί στις προσπάθειες που κάνει η Επίτροπος, δύσκολα μπορώ να φανταστώ πώς το Συμβούλιο θα συμπεριλάβει και αυτά, αυτά τα κριτήρια στο μηχανισμό του Σέγγεν. Πρέπει να σεβαστούμε την ελεύθερη κυκλοφορία των πολιτών και των κεφαλαίων. Αυτό βρίσκεται στη συνείδησή μας και στη συνείδηση όλων. Ο κύριος Έλσιου. Σας ευχαριστώ και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω την νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις λεπτομέρειες την καταλεπτή αυτή ε, γνωμοδότηση. Θα δούμε αν θα ληφθεί υπόψη από το Συμβούλιο ή όχι και θα γίνει δεκτή. Το ελπίζω και εγώ αναφέρομαι στην νομική βάση. Είναι σαφές ότι από την άποψη της νομικής υπηρεσίας το άρθρο 70 μπορεί μόνο να εφαρμόζεται σε περίπτωση που η αξιολόγηση θα γινόταν από τα κράτη-μέλη όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Η ουσία όμως του νέου μηχανισμού που προτείνεται είναι ότι θα παρέχει μια ευρωπαϊκή αξιολόγηση μηχανισμό, όπου θα έχουμε έναν μηχανισμό ευρωπαϊκής αξιολόγησης, όπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι αρμόδια και υπεύθυνη για αυτό το μηχανισμό. Φυσικά υπό τον έλεγχο μιας ε, επιτροπής ε, υπό τη σύνθεση και εκπροσώπηση των κρατών μελών. Πιστεύω ότι ήταν απαράδεκτο αυτό το οποίο συνέβη σε σχέση με, την, ε, με το Συμβούλιο. Πρέπει να αποτροχοποιηθεί, να απελευθερωθεί η κατάσταση όσο των δυνατόν γοργότερα για το νέο μηχανισμό αξιολογήση του Σέγγεν. Διαφορετικά θα υπονομεύσει το Συμβούλιο τα ίδια αυθεντικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει ένα βελτιωμένο σύστημα ε, διαχείριση των εξωτερικών συνόρων και μια καλή διαχείριση και διακυβέρνηση του χώρου Σέγγεν. Όσον αφορά την ε, διαφθορά και το οργανωμένο έγκλημα, Συμμερίζομαι την άποψη που εκφράστηκε από την νομική υπηρεσία. Δηλαδή ότι δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στο φάσμα, στο πλαίσιο της ε, εντολής για το, Schengen, το κοινοτικό κεκτημένο του Σέγγεν. Ο τρόπος φυσικά που το διατυπώνει η νομική υπηρεσία του Ευρωκοινοβουλίου αφήνει εναλλακτικέ δυνατότητες που μπορούν να ληφθούν υπόψη σε περίπτωση αξιολογήσεων επιτόπου ως συμπληρωματικών, παραπληρωματικών, συνοδευτικών μέτρων. Και πάλι για άλλη μια φορά <clears throat> τονίζω θέλω να ξαναπώ ότι είναι δύσκολο να εφαρμοστεί με αυτόν τον τρόπο όπως προτάθηκε η νομική βάση. Χρειάζεται μια αξιολόγηση με αντικειμενικό τρόπο και αντικειμενική βάση. Κανείς δεν μπορεί να αντικειμενικά να μετρήσει την διαφθορά. Αυτό θα οδηγούσε σε υπερβολική γραφειοκρατική επιβάρυνση όσον αφορά τη δράση μας. Πράγμα το οποίο δεν έχει καμιά σχέση ούτε με το εκτιμένο του Σέγγεν ούτε με τις διατάξεις των συνθήκων. Και αυτό καταδεικνύεται τώρα πλέον με κάθε σαφήνεια και το γεγονός ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία δεν κατάφεραν να ενταχθούν στο χώρο Σέγγεν παρότι υλοποιούσαν όλες τις προϋποθέσεις γι' αυτό. Σας ευχαριστώ. Η κυρία Λάτφορντ τώρα έχει τον λόγο παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Εγώ υποστηρίζω απόλυτα αυτά τα οποία ο κύριος Κοέλιο προηγούμενα ανέφερε και στο έργο που επετέλεσε τον υποστηρίζω για αυτή την πρόταση απόλυτα υποστηρίζω, πρέπει να πω, τα επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν από την νομική υπηρεσία και είναι ισχυρά για το ότι η νομική βάση θα πρέπει να είναι το άρθρο 77, προφανώς με συναπόφαση, και ότι ένας κοινοτικό μηχανισμός θα είναι αυτός που θα λειτουργεί, για τον οποίο δεν επαρκεί και δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 70. Επίσης, εκτιμώ το έργο που έχει επιτελέσει μέχρι σήμερα ο Κάρλος Κοέλιο προσπαθώντας να διασφαλίσει τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Ιρλανδία. δεν είναι μία μονομερή τοποθέτηση σε αυτή την ε, αναγνώριση. Είπε και ο Σπέρι, όταν δεν συμμετέχουν δεν μπορεί κανεί να αξιολογήσει τις δικές τους επιδόσεις και ικανότητες όσον αφορά τα θέματα αυτά για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τη συνεργασία των αστυνομικών των διοκτικών αρχών. Και είναι σημαντικό αυτό σε σχέση με την προστασία των, για παράδειγμα, προσωπικών δεδομένων όσον αφορά το Ηνωμένο Βασίλειο. Θα ήθελα, και εδώ πρέπει να το πω αυτό κύριε Κοέλιο, σε σχέση με το Σέγγεν τα βρίσκω μια πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπιστεί για να κατανοήσουμε με σωστό τρόπο τα στοιχεία αυτά για το, τα θέματα αυτά τα οποία με απασχολούν το Ηνωμένο Βασίλειο περιπλέκει το θέμα, περιπλέκει η θέση του το θέμα της συμμετοχής στο Σέγγεν θεωρώ ότι με την, τις δημιουργικές δυνάμεις που υπάρχουν σε σχέση με τους νομοθέτες και τις ε, νομικές υπηρεσίες των τριών θεσμικών οργάνων σίγουρα θα έπρεπε να είναι δυνατό να εξευρεθεί μια διατύπωση, μια πρόταση που θα επιτρέπει την εν μέρη μερική συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και, του Ιρλαν... και της Ιρλανδίας μέσα στο πλαίσιο των ε, δράσεων για το κεκτημένο του Σέγγεν τουλάχιστον. Δεν κατανοώ απόλυτα όλα αυτά τα οποία λέει η νομική υπηρεσία. Σε σχέση με την τελευταία της, τελευταία της γνωμοδότηση διατυπώνει και λέει ότι θα έπρεπε να υπήρχε μια ένα ξεχωριστό νομικό, νομοθετικό ή νομικό μέσο για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας, το ΧΑΣΑΠ που είναι αυτό, και αναφέρονται στη γνωμοδότησή τους πριν από ένα χρόνο για την ε, υπηρεσία ITI και αφορά το IT, την υπηρεσία του IT, μια στιγμή το έχω χάσει αυτή τη στιγμή, που πρότεινε ένα κανονισμό που θα θέσπιζε αυτό τον οργανισμό και μετά τα μέσα για την εντολή που θα αναλάμβανε και για τη διαχείριση για κάθε σύστημα ή κάθε επιμέρους IT θέμα αυτή οργάνωση, αυτός ο οργανισμός. Θεωρούν ότι ακολουθήθηκαν όλα αυτά στον κανονισμό που συγκρότησε και θέσπισε τον οργανισμό της IT, διότι από ό,τι γνωρίζω και είμαι σε θέση να πω, νομίζω ότι μόνο στις αιτιολογικές σκέψεις αναφέρονται το, αναφέρεται το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο συμμετέχει λόγω αυτής, για αυτή την απόφαση και λόγω μιας απόφασης Συμβουλίου μετά από αίτημα του Ηνωμένου Βασιλείου σε σχέση με το άρθρο 4 όσον αφορά το 19 και όσον αφορά τη Eurodac και τις συναφείς δράσεις δεν είναι απόλυτα σαφές από τη διατύπωση αυτή που υπάρχει για το κείμενο για την IT αν ανταποκρίνεται στις απαιτήσει που είχε διατυπώσει η νομική υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν ένα χρόνο για μια ξεχωριστή, για ένα ξεχωριστό όργανο και εδώ πάλι θα ήθελα την κατεύθυνσή σας, την ε, συμβουλή σας σε σχέση με το ερώτημα του κ. Κουέλιο. Τι θα κάνουμε με τη συμμετοχή ε, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας αν ε, δεν είναι δυνατόν με αυτό το, μέσα σε αυτό το πλαίσιο να γίνει και πρέπει να εξευρεθεί μια βάση. Στο πλαίσιο του 77 θα γίνει ή πώς. Η κυρία Ντανόκα παρακαλώ. Yes, thank you, Chair. Θα σε ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομη. Ε, και θα είμαι σύντομη και σε σχέση με αυτή τη γνωμοδότηση ευχαριστώ για την παρουσίασή της, ιδιαίτερα ενθαρρυντική είναι η δήλωση και της Προεδρίας που ανέφερε ότι σε σχέση με την αλλαγή της νομικής βάσης ότι υπάρχει ελπίδα ότι θα υπάρξουν νέα στοιχεία από το, από το Συμβούλιο και από την Πολωνική Προεδρία που θα δείχνουν ότι θα επιληθεί το πρόβλημα. Κάθε επιτυχία στον εισηγητή κύριο Κουέλιο. Είχε υπάρξει η δέσμευση για τροπολογίες για τη 34, 43 και 31. Δεν είμαστε εμείς εκείνοι που καταθέσαμε αυτές τις τροπολογίες, όμως Εν πάση περιπτώσει θα ήθελα να υπογραμμίσω το γεγονός ότι αφορούν την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος όσον αφορά ακριβώς τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Και υπάρχει πραγματική ανάγκη να τονιστεί αυτή η πτυχή, διότι υπάρχουν πολλές εικασίες ότι χρησιμοποιείται αυτό ως μέσο η, ε, ως εργαλείο για την παραβίαση του κεκτημένου του Σέγγεν. Παράδειγμα, σε σχέση με την Νορβηγία κάποιες προαναγγελίες υπήρξαν για πρωτοβουλίες για την εισαγωγή ελέγχων στα σύνορα. Ακριβώς λέει επειδή υπάρχει οργανωμένο έγκλημα από την δική μου χώρα, από την Λετωνία που εισάγεται και περνά στην Νορβηγία. Γι' αυτό λοιπόν σε σχέση με αυτή την αξιολόγηση και σε σχέση με τα έγγραφα, τα έντυπα τα οποία συζητούμε τώρα και τις προτάσεις, ένα πολιτικό μήνυμα είναι αυτό το οποίο αποστέλλεται και είναι αυτό τώρα εκείνο το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να το στείλουμε εμεί ω Ευρωκοινοβούλιο ένα πολιτικό μήνυμα. Πρέπει να είναι α, μια φορά να σαφινιστή ότι το Σέγγεν είναι κάτι που δεν μπορούμε με εικασίες και φήμες ή για κάποιους ιδιωτελείς πολιτικούς σκοπούς να χρησιμοποιήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Έρνστ παρακαλώ. Μάλιστα, σας ευχαριστώ. Πολλά σημαντικά έχουν αναφερθεί, όμως παρόλα αυτά οι ευχαριστίες μου στην νομική υπηρεσία για αυτή την παρουσίαση των προβλημάτων και την νομική γνωμοδότηση. Με καθησυχάζει κάπως και ξέρω γιατί βρίσκομαι εδώ στην Ευρωβουλή και δεν είμαι μάταια εδώ, δεν ματαιοπονώ, δεν πάει του κάκου η παρουσία μου. Η σωστή διαδικασία αξιολόγηση για το Σέγγεν είναι αναπόφευκτο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει, να εμπλέκεται και να είναι ένας κύριος ε, παίκτη στο παιχνίδι. Για το άρθρο για το 77 πρέπει να είναι σαφές και να δώσουμε συνέχεια στην σωστή νομική βάση. Δεύτερο στοιχείο, σύντομα, διαφθορά και καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Όλα πάλι αναφέρθηκαν εδώ. Φυσικά δεν έχει καμιά θέση αυτό εδώ, αυτή η στόχη εδώ. Υπάρχουν και άλλοι λόγοι, το ανέφεραν προλαλήσαντες και έχει αποσαφινιστεί. Ούτε λοιπόν θα επεκταθώ περαιτέρω σε αυτό το σημείο. Με καθησυχάζουν όλα αυτά διότι κατά τα άλλα θα είχαμε κάποια χαοτική κατάσταση, διαφορετικές προδιαγραφές και διατάξεις που θα έπρεπε σε κάθε περίπτωση με διαφορετικό τρόπο να αντιμετωπίζονται και να ισχύουν. Το τρίτο σημείο φυσικά είναι η ενίσχυση, η ενδυνάμωση της διαφάνειας και του ρόλου του Ευρωκοινοβουλίου. Αν δείτε τις τροπολογίες μας και τροπολογίες άλλων, θα διαπιστώσετε ότι εμείς σε όλα τα θέματα θέλουμε το Ευρωκοινοβούλιο να εμπλέκεται, να συμμετέχει και να έχει καθοριστικό ρόλο. Και όταν πρόκειται για τα πολιετή προγράμματα με συστάσεις για τις Φυσικά επιθυμούμε να γνωρίζει εκ προημίου το Κοινοβούλιο για τέτοιε δράσεις και να συμμετέχει και να συνεμπλέκεται. Και πολλά άλλα παρόμοια και στρέφομαι προς τον εισηγητή. Είναι πολύ σημαντικές τέτοιε τροπολογίε και πρέπει να ληφθούν αυτά τα αιτήματα υπόψη. Φυσικά τώρα υπάρχουν και επιφυλάξει και αυτά δεν είναι καινούργια πράγματα. Όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία για παράδειγμα αφορούν ελέγχους στα σύνορα, έστω και περιορισμένους για περιορισμένη διάρκεια, μας προβληματίζουν όλα αυτά. Δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι με αυτά τα οποία διατυπώνει ο εισηγητής. Έχω μεγάλες ανησυχίες. Όλα αυτά δεν είναι αρκετά αυστηρά και περιορισμένα στο εύρος τους ώστε να υπάρχουν τέτοιοι έλεγχοι που θα δεχόμαστε. Γι' αυτό έχω καταθέσει την τροπολογία 52 που αποσαφηνίζει τι επιθυμούμε εμείς και που τονίζει ότι θέλουμε να είναι σεβαστή η κατάργηση των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα. Κύριε Κουέλιο, για σας ήταν αυτό, σε εσά στόχευε. Μάλιστα. Κατά τούτο λοιπόν σε αυτό το σημείο μπορούμε να συζητήσουμε ευρύτερα και σε βάθος αν επιθυμούμε ή όχι ελέγχο στα σύνορα. Έχουμε επιφυλάξει εμείς. Δεν θέλουμε τέτοιους ελέγχους. Επαρκούμε σε αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν τελειώνει εδώ το θέμα αυτό όμως. Ακούσατε κάποιες παρατηρήσεις. Μήπως θέλετε να συνοψίσετε κύριε Κοέλιο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, όλους όσους πήραν το, λόγο για τα σχόλια και τις απόψεις που εξέφρασαν. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό που είπε η Πολωνική Προεδρία. Όταν μας είπαν ότι προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να συμπεριλάβουν το πρώτο και το δεύτερο τμήμα της εντολής ε, ε, της αξιολόγησης του Σέγγεν στο ίδιο μέσο. Είναι κάτι το οποίο ζητούμε από την αρχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, καταπολεμήσαμε τα δύο μέτρα και σταθμά. Είπαμε ότι ο μηχανισμός πρέπει να είναι ένας και ότι οι όροι που θα έπρεπε να επιβάλλονται είτε ε, και για τους όρους για τους οποίους θα έπρεπε να ισχύουν, είτε για, τους, ε, για τα υποψήφια κρατημέλη, είτε για τα ήδη μέλη του Σέγγεν. Ε, βλέπω λοιπόν ότι η Πολωνική Προεδρία ε, θέλει να συμπεριλάβει και το πρώτο και το δεύτερο τμήμα στον ίδιο μηχανισμό. Είναι κάτι που μας ικανοποιεί, μας βρίσκει σύμφωνους και κατά τη γνώμη μου είναι κάτι το οποίο επιτρέπεται στο πλαίσιο της συναπόφασης με το Κοινοβούλιο και ε, στο πλαίσιο του άρθρου 77 συνεπώς. Θα ήθελα να απαντήσω στα σχόλια που έγιναν κύριε Πρόεδρε λέγοντας τα εξής. Πρώτον, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε τον ε, υπάρχοντα μηχανισμό αξιολόγησης, ε, καθιστώντας τον ένα ευρωπαϊκό σύστημα και όχι διακυβερνητικό σύστημα. Δεύτερον, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση με αποτελεσματικό, με αποδοτικό τρόπο. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δεν ισχύει τώρα και όλοι το γνωρίζουμε. Τρίτον, Θέλουμε να βοηθήσουμε τα κράτη-μέλη που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα σε αρκετά πρώιμο στάδιο να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες τους με ενισχυμένο ρόλο της Frontex από πλευράς υποστήριξης. Επίσης θέλουμε να υπάρξουν κυρώσεις σε περίπτωση που ε, εξακολουθούν να υφίστανται οι αδυναμίες και αν ε, θέτουν ένα αμφιβόλο την ε, συνολική ασφάλεια της ζώνης Schengen. Αυτό προσπαθούμε να χτίσουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα διαφορετικό από αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και γι' αυτό το λόγο το Συμβούλιο πρέπει να κάνει μια επιλογή. Ή θα το κάνει αυτό με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή χωρίς και ενάντια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να λάβει την απόφαση αν θέλουν να παραμείνουν με τον ε, ε, μηχανισμό των ισχύοντα ή αν θέλουν να τον τροποποιήσουν, να τον βελτιώσουν, ε, να τον καταστήσουν έναν ευρωπαϊκό μηχανισμό όπως εμείς προσπαθούμε να προτείνουμε. Αυτό επαφίεται στο Συμβούλιο. Αυτό θα λάβει την απόφαση. Από πολιτικής απόψεως, από νομικής απόψεως είναι σαφής η κατάσταση. Αλλά είναι μια πολιτική απόφαση την οποία πρέπει να λάβει το Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα, ευχαριστούμε τον κύριο Κουέλιο, ευχαριστούμε όλους όσους συμμετείχαν ε, στη συζήτηση, τη νομική υπηρεσία για τη γνωμοδότησή της, η οποία επιβεβαιώνει σε αυτό το ε, στάδιο, επιβεβαιώνει και εδρεώνει τη θέση ε, την οποία έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξ αρχής. Νομίζω τώρα ότι είναι η στιγμή να σας αναφέρω ότι θα γίνει μία ψήφος, ε, μία ψηφοφορία προς ανατολισμού το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο του 2011 στην Επιτροπή μας. Έχουμε λοιπόν χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας. Και φτάνουμε στα διάφορα έτσι. Υποθέτω ότι δεν υπάρχουν διάφορα για σήμερα. Καλά τα πήγαμε για σήμερα και θα ήθελα να αναφέρω την επόμενη συνεδρίασή μας ε, που θα λάβει χώρα τον Αύγουστο στις, 21, στις, στις 31 ε, Αυγούστου, διορθώνει ο Πρόεδρος, στις 31 Αυγούστου, 9 η ώρα το πρωί, 9 με 12.30. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Ε, το μόνο που μένει είναι να σας, να σας ευχηθώ καλές ε, διακοπές, καλές καλοκαιρινές διακοπές. Ελπίζω να τα περάσετε πολύ καλά και θα τα ξαναπούμε στις 31 Αυγούστου. Γεια σας.